Καλημέρα σας. Ξέρω ότι πολλοί έχετε πάει και σε προηγούμενη πιο πρωινή ακόμα συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τον ενθουσιασμό σας. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν δύο διαφορές τη γνωμοδότηση για το refit και το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου κ. Γιακοντσάρη. Και έχουν μετακινηθεί και τα δύο θέματα στην επόμενη συνάντησή μας, συνεδρίασή μας. Άρα περνάμε στο 6. Ήταν 6 και τώρα θα γίνουν τα επόμενα θέματα θα πάρουν μικρότερο αριθμό προτεραιότητας. Λοιπόν, ή αύξοντα αριθμό. Ανακοινώσεις. Υπάρχει αναμετάδοση, προσέχετε. Υπάρχει και το e-meeting ή τα συνεδρίαση. <laughs> Υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής των τροπολογιών να μην σημάνει αυτό παρακαλώ ότι θα στείλετε ακόμα περισσότερες τροπολογίες γιατί δεν θέλουμε μόνο ποσότητα αλλά και ποιότητα. Είναι βέβαια ακόμη δοκιμαστικό θα δούμε. Έχουμε και δύο νέα μέλη της γραμματείας. Τον Πίτερ Τραν που απουσιάζει έχει επιστρέψει από πεντάμινη μετάθεση στο Συμβούλιο. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν και θέλουμε να δούμε και τι έμαθε εκεί όταν επιστρέψει. Και την Παρασκευή Ζαβάκη που είναι νέα διοικητική υπάλληλο. Ορίστε εκεί, ευχαριστώ που ήρθατε να μας βοηθήσετε. Και ευχαριστούμε και αποχαιρετίζουμε την Ιωάννα Παππού EPRS, um, growing and again the... που πήγε στο EPRS. Um, now, first, uh, main item. Um, Birgit, would you like to give an update? Θέλει κανείς να μας κάνει μια ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο της περασμένης νύχτας. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χτες το βράδυ είχαμε το πρώτο τριμερή διάλογο για την οδηγία για τα πακέτα, τα ταξιδιωτικά. Πάρα πολύ ε, επικοδομητικός ο διάλογος, η ατμόσφαιρα πάρα πολύ φιλική και ευχάριστη, αλλά και σε πολλά σημεία πρέπει να σας πω συμφωνούμε, αλλά σε αυτά που δεν συμφωνούμε απέχουμε έτη φωτός. Το σημαντικότερο είναι το πεδίο εφαρμογή και ο ορισμός των πακέτων αυτών των ταξιδιωτικών και των ρυθμίσεων που συνδέονται για τις τιμές. Το Συμβούλιο είπε ότι γενικά κάνει μια διάκριση ε, μόνο μεταξύ δύο κατηγοριών. Ε, είτε ε, είναι ε, πακέτο ε, το, η προσφορά είτε είναι ένα ταξίδι με το οποίο συνδέονται κάποιες ε, ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Αλλά το θέμα δεν έχει λυθεί σε καμία περίπτωση από τη προστασία του καταναλωτή και αστικής ευθύνης. από την παλιά οδηγία δεν καλύπτονται οι παροχές υπηρεσιών και ε, οι κρατήσεις από το διαδίκτυο. Ε, είχε κάτι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο το απορρίπτει ως πολύ περίπλοκο. Και έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να το πω κάπως προσεκτικά. Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι αυτό που ζητάμε, ε, τα στοιχεία τα προσωπικά, αριθμός διαβατηρίου και άλλα τέτοια δεδομένα, δεν είναι τμήμα της οδηγίας. Αν γίνει αυτό, είναι άσκοπος κόπος. Παρακαλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το ξανακοιτάξει και εκεί που έχει την αίσθηση ο καταναλωτής ότι είναι σχετικά τα δεδομένα αυτά και πρέπει να αντιμετωπίζονται, θα πρέπει να έχουμε ενιαία μεταρρύθμιση, για ε, αποζημιώσεις ε, και τα λοιπά που ισχύουν και με τα ταξίδια ε, που αγοράζει σε πακέτο. Επίσης έχουμε διαφορές για την προστασία του καταναλωτή, για την υποχρέωση ενημέρωσης και πληροφόρηση. Αυτά λύνονται. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να καλύπτονται από την οδηγία και να έχουμε μια ποιοτική προστασία. 5 Μαρτίου έχει ε, προγραμματιστεί η επόμενη τριμερή συνάντηση. Την Παρασκευή τώρα έχουμε μια ε, τεχνική συνάντηση σε επίπεδο εργασίας. Μετά όμως επειδή πέφτει Στρασβούργο και Τυρκουάζ εβδομάδα, δεν μας φτάνουν δύο ώρες τούτη την Παρασκευή μέχρι το Μάρτιο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εργαστούμε μεθοδικά. Το Συμβούλιο θέλει να τελειώνει το Μάιο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό, αλλά θα πρέπει να ε, ε, χειριστούμε σωστά τα θέματα και να τα διεκπαιρεώσουμε με αρτιότητα. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συγγήτριά μας έκανε εξαιρετική δουλειά εχθές ε, στον τριμερή διάλογο στη διαπραγματευτική ομάδα εξηγώντα τη θέση του Κοινοβουλίου για να μπορέσει η οδηγία αυτή να ενταχθεί ε, στην ψηφιακή εποχή και να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε τώρα σε άλλες ε, καταστάσεις. Και να μην δημιουργηθούν παραθυράκια και ε, προβλήματα και στρεβλωθεί η αγορά. Πολύ καλή δουλειά, μπράβο και ευχαριστώ και ο επόμενος τριμμένος διάλογος θα είναι εδώ στο Κοινοβούλιο. Μόλις με πληροφορούν ότι δεν υπάρχει διερμηνία στα μαλτέζικα. Oh. Συγγνώμη γι' αυτό. Αρρώστησαν οι μαλτέζοι διερμηνείς. Ε. Ελπίζω να γίνουν καλά σύντομα. Μπορείτε να μιλήσετε μαλτέζικα αλλά όχι να ακούτε. The Επόμενο θέμα στη σε διάταξη. Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων TTIP με συντάκτρια γνωμοδότησης κύρια Ντίτα Σαραντσόβα των Φιλελευθέρων. Ε, ε, ξέρετε το TTIP. Θα δώσω μέσω στο λόγο. Αλλά να σας θυμίσω πρώτα ότι θα έχουμε κοινή δημόσια ακρόαση στις 24 Φεβρουαρίου για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες για την εσωτερική αγορά του TTIP. 10.30 με 12.30 θα γίνει αυτή η ακρόαση και θα επικεντρωθούμε σε δύο τομείς που έχουμε αρμοδιότητα και όπου ήδη έχουμε εκπονήσει προτάσεις. Σίγουρα θα μας τα εξηγήσει η συγκήτρια καλύτερα. Αλλά υποπτεύουμε ότι θέλουμε να έχουμε και περισσότερες δημόσιες συζητήσεις για το TTIP υπό την εξαιρετική της καθοδήγηση. Θα της δώσω μέσα το λόγο, κυρία Χαρανσόβα. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πριν αρχίσω το κύριο θέμα, θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη για το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε στην ΙΜΚΟ για τη γνωμοδότηση. Η ΙΝΤΑ πιέζει όλες τις άλλες επιτροπές να βιαστούν υπέρ του δέοντος. Δεν φορολαβαίνουμε καν να σκεφτούμε τις προτεραιότητές μας. Εγώ ζητώ αναβολή μερικές μέρες που δεν θα έχει επιπτώσεις αρνητικές. Σα ζητώ συγγνώμη λοιπόν, αλλά δεν φταίω εγώ για την πίεση χρόνου. Θα ήθελα λοιπόν να πω στους συντονιστές και τους κοιόδης ότι το TTIP θα παραμείνει στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεών μας και μετά την έγκριση αυτής της γνωμοδότησης και γι' αυτό προτείνω να συνεχίσουμε και εμείς να καλούμε την Κομισιόν να έρχεται είτε στην πλήρη επιτροπή είτε στις ομάδες εργασίας για να συζητάμε αυτό το θέμα. Ήδη το πρωί έγινε η πρώτη συζήτηση με τον κύριο διαπραγματευτή και τους κοιόδης. Δεν υπάρχει λόγος να μην συνεχίσουν τέτοιες επαφές μέχρι την τελική έγκριση ψηφοφορία. Εν τω μεταξύ ελπίζω να μπορέσουμε να οργανώσουμε όσο δυνατόν περισσότερες συναντήσεις με τους κοιόδης και τους διαπραγματευτές. Θα ήθελα τώρα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι κάθε ευρωβουλευτής έχει τώρα πρόσβαση στα έγγραφα στο λεγόμενο reading room και έχουν δημοσιευτεί πολλά έγγραφα και online που μπορούν να τα συμβουλευτούν και απλοί πολίτες. Για την ίδια τη γνωμοδότηση τώρα ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι η γνωμοδότηση πρέπει να βασίζεται σε θέματα που εμπίπτουν στις δικαιοδοσίες της Επιτροπής μας. Γι' αυτό στο σχέδιό μου ακολουθώ τη δομή της κύριας έκθεσης αλλά τονίζω μόνο τα θέματα που μας αφορούν. Το TTIP όπως ξέρετε αφορά την ενιαία αγορά και εμάς περισσότερο αφορά αυτό το θέμα. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτά που μας είπε το πρωί ο κύριος διαπραγματευτής. Το ζωτικό θέμα των διαπραγματεύσεων αφορά τις δικαιοδοσίες της ΙΜΚΟ η ελεύθερη διακίνηση αγαθών, τεχνικές προδιαγραφές, δικαίωμα εγκατάστασης, ελευθερία χορήγηση υπηρεσιών, δημόσιες προμήθειες, δυσμιστικά θέματα. Όλα από αυτά θα συζητηθούν και από το TTIP. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ζωτικό η ΙΜΚΟ να παίξει κύριο ρόλο εδώ για το TTIP. Προσωπικά πιστεύω ότι το TTIP εάν γίνει σωστά θα υποβοηθήσει την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Και τα ευρωπαϊκά πρότυπα μπορούν να καταστούν παγκόσμια. Παγκόσμια. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία αναθέρμανσης της εμπιστοσύνης από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το ανέλαβα και προσβλέπω στις πολλές τροπολογίες που θα ενδυναμώσουν το κείμενό μας για όλα αυτά τα θέματα και υποφελεί διάλογο με τους ποιόδης. Σας κατευχαριστώ. Και εμείς σας κατευχαριστούμε πιο πολύ. Ξέρουμε ότι ο καθένας έχει περιορισμό στις γνωμοδοτήσεις και περιορισμένο χρόνο. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Πράγματι νομίζω θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες. Ο κύριος Σόπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Σφάπ, ε, καταπληκτική η πρόταση της συναδελφού Σαράνσοβα. Νομίζω ότι με βάση αυτή μπορούμε να συζητήσουμε πολύ καλά για τα διάφορα σημεία. Ομολογώ ότι σήμερα εγώ δεν έχω πολύ μεγάλη ιδέα για τις τροπολογίες που θα μπορούσε να κάνει κανείς σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κείμενο, έχει πετύχει από την αρχή. Βεβαίω, τα μεγάλα ζητήματα που κυριαρχούν σε αυτή τη συμφωνία αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στο παρόν σχέδιο γνωμοδότησης και ε, τελικά στην ίντα που είναι η αρμόδια επί της ουσίας ε, υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου. Καλό είναι που έχουμε εμεί την γνωμοδότηση, αλλά μόνο στο τέλος θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αν η συμφωνία αυτή ανταποκρίνεται στις επιθυμίες που εκφράζουμε εμείς και που η Επιτροπή ίντα, επαναλαμβάνω, αρμόδια ε, καθήλυν θα ε, προτείνει. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να αναφέρω τα εξή τέσσερα σημεία. Έχει απολύτως δίκιο η κυρία Σαράνσοβα ότι η δική μας Επιτροπή τελικά θα φυγεί περισσότερο από αυτή τη συμφωνία. Όχι μόνο εμείς δηλαδή και η Επιτροπή Περιβάλλοντος φαντάζομαι, αλλά εμά θα μα αφορά πάρα πολύ στην καθημερινή μα δουλειά. Δεν έχω λοιπόν πρόβλημα να δούμε και να προχωρήσουμε την ρυθμιστική συνεργασία, regulatory cooperation, αλλά να μην υπερβάλλουμε έτσι ώστε να μας δεθούν τα χέρια για την νομοθετική δουλειά. Κάθε πρόταση χρειάζεται... Ε, να μελετηθεί για το τι συνέπειε θα έχει όχι μόνο για την εσωτερική αγορά μας, όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και για τη διατλαντική συνεργασία. Είναι απολύτως θεμητό αυτό και αποδεκτό, αλλά δεν νοείται τελικά να περιορίσουμε εμείς και να επηρεάσουμε ε, εκ των προτέρων την νομοθεσία μας λόγω αυτή της συμφωνίας. Θέλω λίγο να κρούσω τον κόδωνα κινδύνου. Δεύτερον, η επαγγελματική κινητικότητα πρέπει να τονιστεί πάρα πολύ. Στα σημεία 3 και 4 τα αναφέρει άλλωστε η συντάκτρια, αλλά ε, οι διαπραγματεύσει θα είναι πιο δύσκολε και πιο σκληρέ από ό,τι αφήνουν να εννοηθεί οι δύο παράγραφοι. Γιατί αυτέ οι αρμοδιότητε στι ΗΠΑ δεν είναι ομοσπονδιακή αρμοδιότητα τη κεντρική κυβέρνηση, αλλά των επιμέρου πολιτιών. Και επειδή στην Ευρώπη έχουμε και εμεί καταστάσεις που χωλαίνουν, θα χρειαστεί χρόνος. Ε, το πιο δύσκολο είναι στο 5, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ε, υπάρχει η ε, νομοθεσία by American στην Αμερική, να προτιμούν τους Αμερικανούς κατασκευαστές και προϊόντα, αλλά αυτό καλύπτει ένα μικρό τμήμα των συμβάσεων. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερες συμβάσεις δεν γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να ε, προωθήσουμε τα αιτήματά μας γιατί αν δεν ανοίξει αυτή η αγορά για τις δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις δεν θα έχουμε και μεγάλο όφελος ε, από τη συμφωνία αυτή στην δική μας εσωτερική αγορά. Και ένα τέταρτο, να πω ένα ε, θετικό, πολύ θετικό παράδειγμα, ήδη έχω κάνει πολλές εκδηλώσεις για το TTIP και έχουμε ένα μικρό φυλάδιο που λέει ότι από στατιστική σκοπιά οι εξαγωγές της Γερμανίας μπορούν να αυξηθούν κατά 94%. Και ήρθε ε, ένας πολίτης και μου λέει «Μα πάτε καλά κύριε Σφάμπ, 94%». λέει «Δεν είναι δικό μου το νούμερο, δεν το κατέβασα εγώ, το λένε οι στατιστικές». Και μετά ζήτησε το λόγο ένας μικρομεσαίος, ε, όπως λέει το σημείο 12, ε, έχει 12 εργαζομένους, είναι στο μέλλον Δρυμό και έχει 2,5 εκατομμύρια τζίρο ε, το χρόνο. Και λέει έχω τεράστια προβλήματα με το τελωνίο ε, για να εκτελονίζω τα διάφορα εμπορεύματα ένα-ένα ξεχωριστά με ετικέτες και διατυπώσεις και πραγματικά ε, αν αρθούν αυτά τα εμπόδια εγώ σίγουρα θα διπλασιάσω τα κέρδη μου ε, γι' αυτό υποστηρίζω πάρα πολύ τη συντάκτρια της νομοδότησης στην προσπάθειά της. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκέπχαρτ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Σαράνσοβα. Είναι πολύ καλή η βάση συζήτηση, η νομοδότησή της και θα συνεργαστούμε. Εγώ δεν βρήκα τίποτα που να διαφωνώ ε, Υπάρχουν αντιθέτω κάποια πράγματα που δεν λέει γνωμοδότηση και θα ήθελα να τη συμπεριλάβει, γι' αυτό θα κάνω και σχετικέ τροπολογίε. Πολύ φυσιολογικό είναι αυτό. Και αν έχουμε σαφείς κανόνες. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε τι μπορεί να περιλαμβάνει μια συμφωνία και τι περιτεύει. Είναι πολύ σημαντικά όσα αναφέρει η γνωμοδότηση, δεν αντιλέγω. Ε, από την άλλη υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας. Έχετε απολύτως δίκιο κυρία Σαράνσοβα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην καλέσουμε διαπραγματευτές και υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ενημερωθεί το σύνολο της Επιτροπής μας για το πώς βαίνουν οι διαπραγματεύσεις. γιατί θα μας επηρεάσει το TTIP πάρα πολύ και την προστασία καταναλωτών αλλά και την εσωτερική αγορά. Θέματα και τα δύο πολύ σημαντικά για μας. Επιτρέψτε μου να απαριθμίσω μερικά σημεία που θέλω να μας απασχολήσουν σε αυτή τη γνωμοδότηση. Το ένα είναι η παροχή υπηρεσιών και ο ορισμός αυτής. Συμφωνώ πολύ με την κυρία Σαράνσοβα εκεί που λέγει ότι Θέλουμε να προσπαθήσουμε τις κοινωνιοφελείς ε, υπηρεσίες με τον τρόπο που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ και ε, επαυξάνω, αλλά το θέμα είναι πώς ορίζονται αυτές οι υπηρεσίες. Γι' αυτό δεν το βρίσκουμε πουθενά, τον ορισμό επαναλαμβάνω. Και τίστε και το θέμα στις διαπραγματεύσεις, εάν ε, θέλουμε να έχουμε θετικούς και αρνητικούς καταλόγους. Και αυτό τι είναι, για ποιες υπηρεσίες δηλαδή πρόκειται. Και τι καλύπτει αυτή η συμφωνία. Να είναι μεγάλη σαφήνεια, χρειάζεται θετικό κατάλογο να λέμε τι συμπεριλαμβάνει, όχι τι δεν καλύπτει αυτή η συμφωνία, γιατί το δεύτερο είναι επικίνδυνο. Ένα δεύτερο που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις υπηρεσίες είναι το εξής. Θα πρέπει να προσέξουμε στον ορισμό των προδιαγραφών και των προτύπων και της τυποποίησης να μην ε, έχουμε έναν αχταρμά. Γιατί γι' αυτό είναι κίνδυνος. Στην περασμένη θητεία είπαμε εμεί ως Κοινοβούλιο ότι δεν θέλουμε γενική και αόριστη τυποποίηση των υπηρεσιών, διότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όσο και ανέφικτο. Και θα πρέπει να συνεχίζει να κυριαρχεί εδώ η πολιτική, να μην μας ξεφύγει ο έλεγχος. Ε, ε, χρειάζεται οπωσδήποτε σαφήνεια όταν μιλάμε για πρότυπα και τυποποίηση. Τι ακριβώς εννοούμε, ιδιαίτερα στα κατανοητικά αγαθά. Ε, παραμένω στις υπηρεσίες, ζητώ συγγνώμη που επιμένω τόσο πολύ και μακρηγορώ, αλλά και το θέμα είναι πώς θα ανοίξουν ε, ε, οι αγορές ε, με βάση ποιες αρχές για την παροχή υπηρεσιών. Θα θυμάστε σίγουρα αυτό που είχαμε συζητήσει για την οδηγία για τις υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, αυτά που βάλαμε εκεί είναι όταν ανοίγει μια υπηρεσία ισχύει η αρχή της χώρας προορισμού και όχι της χώρας προέλευσης και να μην ε, ανατραπεί αυτό λόγω ατυχήματος ή παραδρομής ή δεν ξέρω προσεξίας γιατί θα έχει επιπτώσεις στην αγορά και στην ποιότητα φυσικά των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κάτι άλλο που μου λείπει λίγο εδώ είναι τα τελωνιακά ζητήματα, εκτός και αν ε, το παρέβλεψα. Α, όχι, λέει customs εδώ, γράφει για τελωνία, αλλά θέλει λίγο περισσότερη εξήγηση αυτό και να εστιάσουμε ενδεχομένω στο εξή. Αν θέλουμε μια τέτοια συμφωνία, TTIP, και, ε, δεν μπορεί να εξαιρείται η ψηφιακή αγορά. Είναι τεράστια η σημασία της Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλές οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που αυτή τη στιγμή κατακλείζουν την ευρωπαϊκή αγορά και καλό θα είναι οι δικές μας νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, να έχουν μια ευκαιρία να ευδοκιμήσουν σε αυτή την αγορά. Χρειάζεται προσοχή αυτό. Πρώτο τελευταίο συνεργασία για τα ρυθμιστικά ζητήματα, τα κανονιστικά και αυτά θα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Να μην απεμπολίσουμε τον έλεγχο η πολιτική. Θα πρέπει η πολιτική να προέχει για την προστασία των καταναλωτών, βελτίωση της βελτίωση των κοινωνικών δικαιωμάτων, βελτίωση τη προστασίας του περιβάλλοντος. Να μην μας ξεφύγουν αυτά, φύγουν από τα χέρια μας και να τα αποφασίζουν κάποιοι άλλοι μέσω στρεβλών κανόνων ή να αμφισβητούνται. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε. Και ένα τελευταίο που θέλω οπωσδήποτε να αναφέρω. Αν και ορισμένοι θα πούν δεν μας αφορά, τι σχέση έχουμε εμείς, θα σας πω τι σχέση έχουμε. Είναι το ESTS, διότι Και βέβαια θα έχει επιπτώσεις αυτό και πολύ μεγάλη στην εσωτερική αγορά ανάλογα με τον τρόπο που θα ρυθμιστεί. Και πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ πώς θα γίνει αυτό. Βλέπετε, είναι εξαιρετική, επαναλαμβάνω, η βάση, ε, η γνωμοδότηση της κυρίας Ράσοβα, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία θα πρέπει να επιμείνουμε. Και ένα συμπέρασμα. Κυρία Σαράνσοβα, συμφωνώ απολύτως με τη δική σας νομοδότηση δεν σημαίνει το τέλος των συζητήσεων αυτό ε, για το TTIP. Θα παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις και τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και όχι οποιασδήποτε. Και σε αντίστοιχη περίπτωση θα πρέπει να έχουμε και ανοιχτή την έκβαση, δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να ε, απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία σε περίπτωση που αντιβαίνει στα δικά μας συμφέροντα. Τα ευρωπαϊκά ευχαριστώ. Ο Ντέμις Ντε Ιόγκ ε, παρευρίσκεται όχι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να πάρω το λόγο μετά την ε, κυρία Γκέπχαρτ και έτυχε πολύ καλά αυτό γιατί συμφωνώ απόλυτα με το συμπέρασμα τη. Αν δεν εκπληρώνονται οι σωστέ προποθέσει, το κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο του. Και θα καταλήξει το συμπέρασμα ότι σε μια φάση που η Ευρώπη δυσκολεύεται να ορίσει την αγορά τη, του δικού τη κανόνε και προσπαθεί να τι ομογενοποιήσει, ενώ υπάρχουν διαφωνίε σε πολλά θέματα όπω τη ε, επανακρατικοποίηση κάποιων στοιχείων, γιατί η Ευρώπη προασπίζεται το κοινό συμφέρον. Σε φάση λοιπόν που η Ευρώπη βρίσκεται ίδια σε κρίση, είναι πολύ επικίνδυνο να διαπραγματευόμαστε με έναν εταίρο, ο οποίο ο ίδιο είναι πολύ αποτελεσματικό. Με την ομοσπονδιακή του διάρθρωση μπορεί να διαπραγματευτεί διαφορετικά του κανόνε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την γνωμοδότηση, ευχαριστώ την εισηγητρία. Όμω, εγώ σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να δω ποιο είναι το πλεονέκτημα και το όφελο για του καταναλωτέ, διότι σε αυτή την επιτροπή πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το, με αυτό το σκέλο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι ωφέλη θα έχουν οι καταναλωτέ από αυτή τη διατλαντική αγορά. Ε, περιμένω όμω, αν θέλετε, να μου το δείξετε και να μου το αποδείξετε. Και θα συμφωνήσω με την κυρία Γκέπχαρτ στο θέμα του SDS. δεν είναι μόνο θέμα της ε, διεθνού ε, αγοράς γιατί είναι το 40% των διεθνών ε, εμπορικών συναλλαγών, είναι τεράστιο όγκο για, για την παγκόσμια αγορά, αλλά θα πρέπει τα κράτη να δίνουν λογαριασμό για τους δημόσιου λογαριασμού, του κατοικούς λογαριασμού, σε ιδιωτικά όργανα επίλυσης διαφορών. Θα είναι πολύ δύσκολο εκεί λοιπόν να υπάρξει ισότητα, διότι οι πολυεθνικέ που βρισκόνται σε μια λογική τη αγορά και έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στην ιδιωτική δικαιοσύνη δεν θα βρίσκονται στην ίδια θέση με τι μικρομεσαίε ή τι μικρότατε επιχειρήσει που θα είναι υποχρεωμένε να συμβαστούν με τι νέε αυτέ συνθήκε. Και θα ε, προσφεύγουν στα κρατικά δικαστήρια. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο μείζον ζήτημα που πρέπει να ε, λυθεί αναφέρθηκε, δεν θέλω να επιμείνω, το θέμα τη ρυθμιστική συνεργασία. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό το θέμα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε την πολιτική κυριαρχία και τι αποφάσει που θα λαμβάνονται από τι εθνικέ βουλέ, τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι πολύ δύσκολο να μην οριστούν σωστά οι όροι τη ε, ρυθμιστικής συνεργασία και επίση κάτι άλλο θα αποτελέσει μέρο τη συζήτηση η διαφύλαξη των κρατικών υπηρεσιών και η πρόσβαση στι δημόσιε προμήθειε. Αυτά πρέπει να ρυθμιστούν. Διότι τώρα στην Ευρώπη έχουμε έναν άνοιγμα προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που είναι πολύ σημαντικά και δύσκολο να τα σεβαστεί κανεί. Εάν αυτά συμπεριληφθούν στην ε, Διατλαντική Συμφωνία, που θα έχουν πολύ μεγάλη νομική βαρύτητα, ε, αυτά πρέπει να συζητηθούν και να ρυθμιστούν εκ των προτέρων. Το συμπέρασμά μου λοιπόν είναι ακριβώ το ίδιο με την κυρία Γκέπχαρτ. Δηλαδή, εάν η Ευρώπη είναι σε θέση να διαφυλάξει αυτά που θεωρεί ουσιαώδη για τη λειτουργία τη, δηλαδή τι κανόνε για την προστασία των καταναλωτών, την υγεία των περιβάλλων, την ε, δικαιοσύνη, του κράτο δικαίου. Εάν αυτά μπορούμε να τα διαφυλάξουμε, τόσο το καλύτερο. Εάν όχι, θα πρέπει να δούμε τι συνέπειε θα υπάρξουν και να λάβει το κοινοβούλιο το ρόλο του. Ευχαριστώ. Έχω έναν μακροσκελή κατάλογο αγορητών, αλλά αν θέλετε κι άλλοι το λόγο, να μα το πείτε. Grappini, Eva Paunova, Catherine Steiler, Marlene Mitzi, and Mylena Trozitsky. And I would like to have a word at the end as well, if I can have a chance. Dan Dalton, Tunisia. Thank you very much. Um, Emma Σας Η κυρία Μακλάρκιν είναι η στιώδης μας, αλλά λείπει και μου ζήτησε να μιλήσω εγώ στη θέση τη εκ των συντηρητικών. Και εμεί ευχαριστούμε για την εισήγηση. Τρία θέματα θέλουμε να θίξουμε εδώ. Πρώτον, το αίτημα να καταργηθούν οι άδειε εργασία. Αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνος γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο το σύστημα λειτουργεί πολύ καλά και είναι ευαίσθητο θέμα. Δεν θέλουμε βέβαια να παρεμποδιστούν οι διαπραγματεύσει του ΤΤΠ με βάση αυτό το θέμα. Τώρα για τη συνεργασία αυτή καλύπτει μόνο προς στιγμή τις κεντρικές κυβερνήσεις και αυτό πρέπει να τονίζεται κρατικό επίπεδο δηλαδή. Όποτε υπάρχουν νομοθεσίες που επηρεάζουν το εμπόριο χρειαπετούν ιδιαίτερη διαφάνεια. θέλουμε σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης οι προμήθειες, ιδίως σε κρατικό και δημοτικό επίπεδο, να σέβονται όσα έχουν συμφωνηθεί για τις δημόσιες προμήθειες. Και φυσικά τα Buy Αμέρικα δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Αν υπάρξει συμφωνία για το TTIP πρέπει να έχουμε μια κοινή αγορά και επί αυτού. Και τέλος, για τους καταναλωτάς. Για μένα το TTIP είναι τεράστια ευκαιρία για τους καταναλωτάς, διότι δίνει τη δυνατότητα να καταργηθούν οι δασμοί. Και αυτό θα ήταν μεγάλη νίκη για τους καταναλωτάς. Φτηνότερα αγαθά, περισσότερη επιλογή. Όλα αυτά σημαίνουν μείωση του κόστου ζωής και αυτό είναι πολύ ζωτικό αν μπορούμε να απαιτήσουμε μια σωστή συμφωνία τίτλου. Μάρκ Ταραμπέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα έλεγα ότι έχω μια θετική προσέγγιση προς την ε, γνωμοδότηση της κυρία ε, Σρέντοβα ε, και πρέπει να πω ότι κάποια από τα σχόλια της κυρίας Γιάννη θα πρέπει να τα δούμε από το φω των εξή τριών σχολείων. Πρώτον, να φροντίσουμε Πώ θα δούμε τι ρυθμίσει. Δεν πρέπει να γίνει ένα επιχείρημα τιμή για μα. Θέλουμε να δοθεί έμφαση στην προστασία των καταναλωτών και υπογραμμίζω τη λέξη αυτή. Αλλά ο στόχο δεν είναι να βρούμε σημεία σύγκληση με τι ΗΠΑ σε διεθνέ επίπεδο που δεν προστατεύουν τόσο καλά του προκαταναλωτέ εμεί. Ούτε θέλουμε μη δημοκρατικά μέτρα για να αποδιαρθρώσουμε κανόνε που πολύ δυσκολία οικοδομήσαμε ω τώρα με δημοκρατικό τρόπο. Επίσης για τις μεγάλες αγορές ε, ένα άνοιγμα σίγουρα το θέλουμε, αλλά εμείς είμαστε οι διεθνείς φορείς της αγοράς, οι διεθνείς παίκτες που περισσότερα από όλους έχουμε ανοίξει τα σύνορά μας. Κάποιοι που δηλώνουν ότι είναι πάρα πολύ φιλελεύθεροι έχουν προστατευτικέ συμπεριφορέ πολύ πιο έντονε από τι δικέ μα. Και δεν θα το εξηγήσουμε αυτό σήμερα. Είναι πολύ έντονο ο προστατευτισμό των ε, Αμερικανών. Και ισχύει και για άλλου ε, διεθνεί ε, φορεί τη αγορά. Γι' αυτό λοιπόν να μην παρασυρθούμε στι δημόσιε ε, αγορέ, τι δημόσιε προμήθειε που αφορούν και τι υποδομέ και τα αγαθά και τις, τα μεγάλα έργα. Και για τον μηχανισμό επίλυση των διαφορών από, από ιδιωτικά όργανα θα πρέπει αυτό να το προσέξουμε επίση. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Διότι οι μηχανισμοί αυτοί υποτίθεται ότι καταπολεμούν ή προστατεύουν μάλλον τις επενδύσεις Καταρχάς, είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να ε, πληγούν οι κανόνες για την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος. Ε, λόγω, να δώσω ένα παράδειγμα. Η κανοβιομηχανία, η Φίλιπ Μόρις στην, ε, στις ΗΠΑ έχει ε, προσφύγει κατά της Αυστραλίας που έχει προσθέσει ένα αυτοκόλλητο στα πακέτα των τσιγάρων για να πει ότι το τσιγάρο βλάπτει σοβαρά την, υγεία. Πολύ συχνά λοιπόν θα μπορεί σε ένα ιδιωτικό δικαστήριο οι πολυεθνικές να προσφύγουν κατά των κρατών, είτε τη ευρωπαϊκή είτε τη αμερικανική δικαιοσύνη, μην ξεχνώντα ότι έχουμε ένα δημόσιο δικαστικό τομέα που είναι πολύ αποτελεσματικό, ενώ με το ιδιωτικό ε, μηχανισμό, με τον ιδιωτικό μηχανισμό επίλυση διαφορών, θα έχουμε ένα μηχανισμό απορδιάρθρωση των κανόνων που έχουμε τώρα. Εδώ λοιπόν ε, αυτέ οι τρει παρατηρήσει για να σα πω ότι σίγουρα θα πρέπει να προσθεθούν τροπολογίε για αυτά τα τρία συγκεκριμένα σημεία. Τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για την έκθεση που με έχει συντάξει. Είναι ένα πολύ χρήσιμο σημείο αφιτηρίας για να δούμε θέματα που αφορούν όχι μόνο την Επιτροπή μας, αλλά μια πολιτική συζήτηση που πρέπει να ξεκινήσουμε και στα επίπεδο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου αλλά και για τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά για τις χώρες μας. Είναι πολύ ε, μεγάλη σημασία. Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αντικειμενικώς είναι μεγάλη μεγάλη ευκαιρία. Και μπορεί να ωφεληθούμε ώστε για την Ευρώπη να προκύψουν νέες εμπορικές ευκαιρίες και η ευρωπαϊκή αγορά να έχει περισσότερες δυνατότητες στην αμερικανική αγορά. Θα πρέπει να πάψουμε να είμαστε τα μικρά αδερφάκια των Ηνωμένων Πολιτειών και να καθόμαστε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες θυμίζοντας ότι έχουμε 500 εκατομμύρια ε, κατοίκους και καταναλωτές ενδεχόμενους περισσότερο από ότι εκείνοι που έχουν 300. Ε, θα έπρεπε εδώ να υπάρχει λοιπόν μια ευρωπαϊκή υπερηφάνεια και με το κεφάλι ψηλά να επιδιώκουμε τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Είναι σημαντικό και αυτό. Νομίζω ότι τα σημεία όπου πρέπει να υπάρξουν βελτιώσει είναι πολλά και διάφορα. Εκεί που θέλουμε να πετύχουμε ευκαιρίε για την Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να ασχολείται με του δασμού, αν και σε πολλά θέματα είναι ήδη χαμηλή και στη ε, μη δασμολογική συνεργασία και τι σχετικέ ρυθμίσει Εδώ Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία όπου η συμφωνία αυτή μπορεί να προσφέρει δυνατότητε στην ευρωπαϊκή αγορά και τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λένε ότι οι ευρωπαϊκέ εταιρείε έχουν κόστο μεγαλύτερο του 10% όπω τον τομέα των αναψυκτικών που φτάνουν στο 70% λόγω των δασμολογικών ε, φραγμών για πρόσβαση στην Αμερικανική αγορά. Ε, σε αυτό τον τομέα, σε αυτού του κλάδου. Πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε κάποιε περαιτέρω διευκολύνσει για τι εταιρείε μα για να ανοίξει και για αυτέ η αγορά και νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξουμε μια συμφωνία που να μην υποβιβάζει αλλά να αυξάνει τι ε, δυνατότητε. Δηλαδή, όταν διαπραγματευόμαστε με τι ΗΠΑ για ρυθμιστικά ζητήματα, είναι πολλέ οι που αφορούν ε, αφορούν ε, πράγματα ίσονο σημασία, Όπω το αν τα φλάστα αυτοκίνητο είναι πορτοκαλί κίτρινα. Αλλά υπάρχουν μεγάλες εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίες ε, που μπορούν να τα καλύψουν αυτά. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή αγορά, αλλά έτσι καλώς αυτές οι εταιρείες έχουν ε, διεθνέ άνοιγμα μπορούν να φροντίσουν τα αυτοκίνητα να είναι ανάλογα με τι απαιτήσει τη μια τη άλλη αγορά. Όμω αυτό που θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία στι επιχειρήσει να ξεπεράσουν τι δασμολογικέ δυσκολίε και του φραγμού. Εκεί πρέπει να κοιτάξουμε να δώσουμε προσοχή και εκεί θα πρέπει να στοχεύσουμε στο να χρησιμοποιηθούν οι καλύτεροι κανόνε για την προστασία των καταναλωτών και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι όλοι οι τομεί, τομεί όπου έχουμε του καλύτερου κανόνε εμεί και προστατεύουμε καλύτερα του καταναλωτέ. Σε μερικέ περιπτώσει οι Αμερικανικοί κανόνε είναι καλύτερα από του Ευρωπαϊκού. Πιστεύω λοιπόν ότι καλό θα ήταν όταν ε, καθίσουμε να αντιπροσωπευτούμε από κοινού να αποφασίσουμε να επιλέξουμε του κανόνε τη μια ή τη άλλη πλευρά που είναι οι καλύτεροι για του καταναλωτέ. Αυτή είναι μια τακτική, ένα κανόνα που θα μα επέβαλε να βελτιώσουμε κάποιου κανόνε υπέρ των καταναλωτών και πολλέ προσαρμογέ θα πετυχθούν και από τι ΗΠΑ. Για τα υγειονομικά και τα φυτογειονομικά λόγω χάρη, η Ευρώπη είναι πολύ πιο μπροστά από τις ΗΠΑ. Αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε ως προβάδισμα. Έπειτα το θέμα των ε, δημοσίων υπηρεσιών. Εκεί από τι διαπραγματεύσεις, πρέπει να αποκλειστούν ε, οπωσδήποτε αυτές, ε, όπως προβλέπει και η δημοτευτική εντολή, και κατέλαβαν εν τέλει είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν ένα σύστημα κανόνων για την προέλευση των προϊόντων που είναι πολύ δυσμευτική και πολύ αυστηρή εδώ και χρόνια. Η Ευρώπη δεν έχει τέτοιους κανόνες. Το Κοινοβούλιο συνεισέφερε στη σχετική συζήτηση, αλλά από αυτού η Ευρώπη θα πρέπει να προσπαθήσει να καταλήξει σε μια θέση λίγο πιο προηγμένη. Όσο για τις προμήθειες, πολλά πράγματα ήδη υπόθηκαν και θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Όμως το τελευταίο που ήθελα να τονίσω, κάτι που απασχολεί πολύ την κοινή γνώμη και το Κοινοβούλιο, είναι το θέμα του μηχανισμού επίλυσης ε, διαφορών μεταξύ κρατών και ιδιωτικών επενδυτών. Εδώ πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία ώστε οι μηχανισμοί αυτοί να δημιουργηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο ώστε να εγγυηθούμε τι επενδύσει, την προστασία των καταναλωτών και ταυτόχρονα να αποφύγουμε τέτοιες ε, πτυχές που μπορεί να ε, περιορίσουν την πολιτική βούληση των κρατών χωρίς να πλήττονται είτε οι επενδύσεις είτε οι καταναλωτές. Όπως είπε και η συγγήτρια, το θέμα αυτό είναι τόσο σημαντικό που θα πρέπει να το δούμε διαρκή και μόνιμη προσοχή από την ε, Επιτροπή μας. Διότι οι επιπτώσεις για την εσωτερική αγορά θα είναι πολύ μεγάλες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Γραπίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να δηλώσω πόσο εκτιμώ το έγγραφο Τζίτα. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά και με την Εύελιν συμφωνώ για τις προσθήκες που ζητάει. Για μας υπάρχουν ακόμα μερικές ασάφειες όμως. Πώς μπορούμε να επηρεάσουμε την Κομισιόν με αυτό το έγγραφο. Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε αλλά θα το ακούσουν ή θα μας αγνοήσουν. Θα λάβουν υπόψη τους τις ανησυχίες και ευχές μας. Εμείς πρέπει να έχουμε τον πρώτο λόγο. Μιλάμε για ενιαία αγορά, για την ευρωπαϊκή αγορά και για σύμβαση με μια άλλη αγορά. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που έχουμε 500 εκατομμύρια καταναλωτάς ενώ εκείνοι μόνο 300. Θα έπρεπε αυτοί να έρχονται εδώ για να ζητήσουν να εκμεταλλευτούν τη τεράστια αγορά μας και δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο που είπε πρέπει να ικανοποιούνται οι καταναλωτές μας γιατί θα είναι φτηνότερα τα προϊόντα. Όχι δεν αρκεί αυτό. Θέλουμε να είναι και ασφαλή και καλύτερης ποιότητας, όχι αναγκαστικά φτηνότερα. Εμείς έχουμε πρότυπα η ευρωπαϊκή αγορά και η αμερικανική αγορά βασίζονται σε διαφορετικά πρότυπα. Εκεί θα υπάρξει το πρόβλημα. Γιατί θα μας κατακλείσουν από παντός είδους προϊόντα χωρίς φραγμούς, χωρίς καμία προστασία και θα λέμε απλώς «Α, τι ωραία θα έχουμε φτηνότερα προϊόντα». Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας και οι βιομηχανίες μας στην Ένωση μπορεί να κινδυνεύουν διότι εδώ δεν βλέπω τίποτα που να φροντίζει τα συμφέροντά τους. Χρειαζόμαστε πολύ στεναρές διαπραγματεύσεις για αυτή τη συνθήκη. Δεν, μπορεί, δεν πρέπει να τυφλωνόμαστε και να ζαλιζόμαστε και να ενθουσιαζόμαστε γιατί θα έχουμε στην προϊόντα. Χρειάζεται ψυχραιμία να τονίσουμε την ασφάλεια, την προστασία των καταναλωτών, την ποιότητα. Ό,τι κάνουμε εδώ στην Ένωση βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια. Θέλουμε οικονομική ανάπτυξη, θέλουμε απασχόληση και αν αποφασίσουμε ότι αυτή η συνθήκη είναι σημαντικότερη από την απασχόληση και την ανάπτυξη θα αποτύχουμε αν θέλουμε απλώς φθηνότερα προϊόντα δεν θα έχουμε εκπληρώσει τους στόχους της δηλωμένης πολιτικής μας. Το, δεν χρειαζόμαστε καθόλου να έρχονται ιδιώτες επενδυτές και να παίρνουν στα δικαστήρια ολόκληρα κράτη με βάση αυτή τη συμφωνία. Εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο και εκείνοι της Κομισιόν που κάνουν τις διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι βέβαιοι ότι ξέρουν ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της συνθήκης. Εύα Πάνοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την εισηγητριά για την πολύ καλή δουλειά της, ε, άριστη για την ακρίβεια. Δύο παρατηρήσει θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα για τις απαιτήσει για τους πολίτες. Εάν θέλουμε να έχουμε ε, μια ενιαία διατλαντική αγορά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την απλή πρόσβαση έροντας τις υπάρχουσες, ε, τους υπάρχοντες περιορισμούς που δυσκολεύουν την κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών και πρέπει να καταργήσουμε τις απαιτήσεις θεωρήσεων για τους πολίτες και τις χώρες που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα διευκόλυνσης θεωρήσεων. Αυτό νομίζω ότι όντως θα επιτρέψει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μεταξύ των ε, εμπορευμένων εταίρων. Το δεύτερο σχόλιο αφορά τα σημεία 12 και 13 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα κεντρικό στοιχείο των συζητήσεων στις διαπραγματεύσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι συναλλαγές τους είναι αυτό που θέλουμε να στηριχθεί στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό για τις μικρομεσαίες πρέπει να δώσουμε έμφαση στις διαπραγματεύσεις από το συμπεριλάβουμε για να καλυφθούν τα εμπορικά συμφέροντα των εταιριών. Δηλαδή, μια πλατφόρμα, ενιαία πλατφόρμα για τα προϊόντα ε, ε, διαδικτυακά και να ενημερώνει τις ρυθμίσεις και τις απαιτήσει δασμολογικού τύπου που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εταιρείε αμερικανικές και ευρωπαϊκές από τη μια την άλλη πλευρά, αλλά και η παρακολούθηση και η υλοποίηση της συμφωνίας θα πρέπει τεχνικώς να λάβουν χώρα με τη συμμετοχή της ε, ε, ε, κοινότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να αποφελούνται πλήρω από του θεσμικού μηχανισμού που θα προκαλέσει και θα οδηγήσει στη δημιουργία του η συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά στοιχεία ήδη καλύφθηκαν, αλλά στην αίθουσα αυτή μόλι, χθε το απόγευμα, είχαμε 200 ακτιβιστέ κατά τη συμφωνία TTIP, που μερικοί ήταν και από την εκλογική μου περιφέρεια στην Σκωτία και ήταν πολύ ενδιαφέρον να του ακούμε, γιατί πολλοί έχουν παραπληροφορηθεί. Έχουν μαθαίνετε ανησυχίε βέβαια. Αλλά υπάρχει πολύ υποψία μεταξύ των πολιτών. Είναι κρίμα για μερικά στοιχεία. Όμω για του διαπραγματευτικού γύρου που έχουν εκπληρωθεί ω τώρα, έτσι κι δεν έχουμε καταλήξει κάτι χειροπιαστό. Οπότε δεν θα πρέπει από τώρα να τα βάζουμε με τον ε, αγγελιοφόρο και να ανησυχούμε για προσωρινές καταστάσεις. Όταν έγινε πριν ένα χρόνο πρώτο πρώτη παρουσίαση σε αυτή την Επιτροπή για τη Συμφωνία TTIP, Λέγαμε ότι θέλουμε να δημιουργηθεί μια κοινή αγορά από τη μια και την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Τεράστιο δυναμικό εφόσον πετύχει και με τι προτεγραφέ που αναφέρει η έκθεση τη εισηγήτρια και τη διατήρηση με την υψηλή ε, προστασία των καταναλωτών όπω την έχουμε στην Ευρώπη, τι υψηλέ απαιτήσει για τα τρόφιμα και το καθεξή. Πρέπει όμω όλα αυτά να γίνουν με τον σωστό τρόπο. Υπάρχουν θέματα διαφάνεια, ξέρουμε ε, ότι πρέπει όλοι να πιστούν, όχι μόνο μερικοί, και οι εθνικές βουλές επίσης να δώσουν το πράσινο φως στο τέλος αυτής της διαδικασίας για να τοποθετηθούν με ένα ναι ή όχι. Και οι παρατηρήσεις που έκανε η κυρία Γκέπχαρτ ήταν σωστές όπως το σημείο 7. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, όπως λέει και η έκθεση αυτή, στο 8 για τα πρώτα και τις προδιαγραφές. Όταν τα είδαμε πριν ένα χρόνο σε αυτή την Επιτροπή, δυστυχώς, τάση να υπάρξει και να δημιουργηθεί ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των φορέων ε, κατάρτισης προτύπων από την Ευρώπη και την Αμερική δεν προχώρησε στο φθινόπορο. Πέρσι μας είχαν πει στην Επιτροπή μας ότι αυτό το μνημόνιο θα είχε προβλεφθεί και τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Πρέπει να πιέσουμε γι' αυτό. Καλά το λέει η έκθεσή σας. Είναι σημαντικό. Πρέπει να προωθηθεί αυτή η προσπάθεια γιατί εάν κερδίσουμε εμπιστοσύνη για τις προδιαγραφές και το υψηλό επίπεδο των προτύπων θα έχουμε ήδη λάβει τη σωστή κατεύθυνση. Στο σημείο 14 για το ελεύθερο εμπόριο. Ήθελα κάποιε αποσαφηνήσει εδώ. Διότι η κατανόησή μου για το ελεύθερο εμπόριο είναι ότι μιλάμε για μια για το δίκαιο εμπόριο θα πρέπει να, για το δίκαιο εμπόριο λοιπόν, για το fair trade, θα πρέπει να το, να το ορίσουμε σε διεθνή επίπεδο και εκεί να υπάρξουν κάποιε αποσαφηνήσει. Θα πρέπει ο διάλογο αυτό να συνεχιστεί, να καλύψουμε τι ανησυχίε των πολιτών και για θέματα όπω οι δημόσιε υπηρεσία, το μηχανισμό επίλυσης ε, μεταξύ κρατών και ιδιωτών επενδυτών. Και αν υπομονώ, να συνεχιστούν αυτές οι εντατικές συζητήσεις που θα έχουμε καθώς προχωρούμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. κυρία Μίτση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολλά από αυτά που θέλω να πω έχουν ήδη Θα συγχαρώ την εισηγητρία, γιατί θεωρώ ότι η έκθεση είναι πολύ καλή. Και πρέπει να πω ότι με την Εύελιν και τη Μαρία Συμφωνούμε ότι αυτή η συμφωνία θα υποφελήσει, θα την Ευρώπη, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, του καταναλωτέ και, και του ε, εμπορευόμενου, εάν οι διαπραγματεύσει οργανωθούν σωστά. Η διαφάνεια λοιπόν εδώ είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν θέλουμε να έχουμε αντιδράσει και διαμαρτυρίε εδώ. Θα πρέπει να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο προστασία τη Ευρώπη. Και ανησυχώ με τον ενθουσιασμό που δείχνουν κάποιοι ότι θα έχουμε τόσο φθηνότερα προϊόντα εδώ στην Ευρώπη και οι καταναλωτέ θα καταχαρούν. Ε, μην ξεχνάμε ότι οι καταναλωτέ θα χαρούν με τι ε, χαμηλότερε τιμέ, αλλά όχι ει βάρο ε, τη απώλεια, ει βάρο των θέσεων εργασία, διότι είναι πολλέ εταιρείε που λειτουργούν εδώ αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εάν χαθούν δουλειέ, δεν θα μπορούν να καν να αγοράσουν τα υπέροχα αυτήνα προϊόντα των Αμερικανών οι Ευρωπαίοι. Πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε το πολιτικό πεδίο, τον πολιτικό χαρακτήρα και τον οικονομικό χαρακτήρα αυτή τη συμφωνία. Δεν είμαι βέβαιο ότι συνδυάζονται, γι' αυτό πρέπει να είναι το επίπεδο επιφυλακή μα πολύ ψηλό. Ιδίω Ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Να μην ωφελήσουμε δηλαδή κάποιον από του φορεί τη αγορά ει βάρο κάποιου άλλου. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί με το πώ θα επηρεαστούν όλοι οι προηγούμενοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει η κατάσταση να αποφέρει ωφέλη και για τις δύο πλευρές, δηλαδή για την Ευρώπη. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι είμαι κατά τη συμφωνία αυτή. Το αντίθετο. Ε, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλες οι ευκαιρίες και όλες οι προκλήσεις που προκύπτουν με την δημιουργία μιας τέσσερα τεράστια αγοράς δεν θα μας παρασύρει. Δεν είναι καλή ιδέα να τα πετάξουμε όλα στο καλάθι των αχρήστων μαζί, αλλά καλό είναι να βγει η Ευρώπη ωφελημένη από όλες τις ε, οπτικέ γωνίες. Ε, οι καταναλωτέ, οι εταιρείε και οι μικρομεσαίες που είναι η ραχοκαλιά της Ευρώπης. Κάτι που είναι μικρό για τις ΗΠΑ τη διαστάσεις του, δεν σημαίνει ότι είναι μικρό και για την Ευρώπη. Α βεβαιωθούμε λοιπόν για το εξή σημαντικό, να υπάρξει διαφάνεια και η Κάθριν τόνισε ότι ε, υπάρχουν ε, πολλοί ακτιβιστέ που τοποθετούνται κατά τη συμφωνία TTIP και έχουν και δίκιο γιατί μερικέ φορέ δεν πληροφορούνται σωστά. Πάρα πληροφορούνται. Έχουμε λοιπόν καθήκον προ του 500 εκατομμύρια ε, πολίτε, οι οποίοι δεν πρέπει όλοι να παραπληροφορηθούν, να προσέξουμε λοιπόν τη διαφάνεια και να υπάρξει δίκαιη διπλωμάτευση. Η κυρία Τραζίνσκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα κάποιους από εσά προηγουμένως να λένε πώς θα οργανωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις και κυρίως πώς θα συνεννοηθούμε με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ε, κάποιοι παραπονέθηκαν ότι άλλες επιτροπές ε, εκτός από το αυτή του Διεθνούς Εμπορίου θα πρέπει να αναλάβουν για την συμφωνία αυτή. Να θυμίσω ότι η πρώτη υπεύθυνη για την συμφωνία αυτή είναι η ευρωπαϊκή Λαή και τα 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Τώρα για το σχέδιο γνωμοδότησης που κοιτάζουμε και εξετάζουμε στην Επιτροπή ΙΝΤΑ να πω ότι υπάρχουν και εκεί αμφιβολίες για τη συμφωνία αυτή, όμως επειδή θέλει τεράστιος ο αντίκτυπος ε, της συμφωνίας αυτής για την καθημερινότητα των Ευρωπαίων, που εσείς προσωπείτε εδώ, και που ε, σε μεγάλο βαθμό μάλλον διαφωνούν, θα έλεγα ότι έχουμε ακολουθήσει μια στάση αφελή και επικίνδυνη. Διότι υπάρχει εδώ κίνδυνο και απειλή για την ε, κυριαρχία των ευρωπαϊκών κρατών και την προστασία των καταναλωτών. Ακόμη και κάποιε ανησυχίε δειλά έχουν εκφραστεί και προθεθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως από τα μέλη της Επιτροπής ΙΝΤΑ, για την ισοπαίδωση των ευρωπαϊκών κανόνων, για την ιδιωτική δικαιοσύνη που θα χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις ε, που χρειάζεται διατησία και για την υλοποίηση, την αδιαφανή υλοποίηση αυτής της συνθήκης. Εγώ παραμένω επιφυλακτική με τη στάση του Κοινοβουλίου ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις ΗΠΑ. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε τα γρανάζια της παγκοσμιοποίησης που μας οδηγούν σε χρονοβόρες διαδικασίες για να δημιουργηθεί μια τεράστια κοινή αγορά με την εμπορευματοποίηση του ίδιου μα του πληθυσμού. δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι συμφωνώ το περιεχόμενο τη ε, γνωμοδότησή σα, όσο και αν είστε υπέρ τη Ευρώπη, διότι οι συγκεκριμένε συστάσει προβλέπουν κάποιε επιπτώσει δεδομένε για τη ζωή των συμπατριωτών μα. Με την συμφωνία αυτή ε, θα πάμε, να χτυπήσουμε με το κεφάλι σε τείχο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και μερικέ σκέψεις από πλευρά μου τώρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η γνωμοδότηση τη ηγητρίας, ιδιαίτερα εκεί που λέει ότι είναι μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθούν πρότυπα και νόμοι υψηλή ε, ποιότητας για τους καταναλωτές και θα είναι διεθνή πρότυπα. Εγώ θα έλεγα μάλιστα παγκόσμια, όχι απλώ διεθνή. Είναι μοναδική ευκαιρία αυτή να έχουμε υψηλέ προδιαγραφές για τους καταναλωτές και μάλιστα όχι μόνο στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο. Δεν συμφωνούμε πάντα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε μια νέα προσέγγιση για να περάσουμε σε παγκόσμια πρότυπα. Είναι πραγματικά μοναδική ευκαιρία και θα πρέπει οπωσδήποτε να διαμορφώσουμε έτσι την συμφωνία ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε και όχι να την απορρίπτουμε από χέρι πριν αρχίσει η διαπραγμάτευση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ωφέλη και τα ευεργετήματα για τους καταναλωτές, είναι σημαντική η οικονομία και η αξία που έχουμε από την ε, άρση των φραγμών δασμολογικών και άλλων. Υπάρχει κόσμος που δεν το βγάζει πέρα. Δηλαδή ε, αν μειωθούν οι τιμές κατά 20% στα τρόφιμα, ας πούμε 10% στα αυτοκίνητα, αυτό είναι σημαντικό όφελος για πολλούς καταναλωτές. Αλλά δεν θα πρέπει να χαθούν θέσει εργασία και ο Νικολοντάντε και ο Ανδρέα Σβάπ έδωσαν παραδείγματα για επιχειρήσεις που βλέπουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα από αυτό το εμπόριο. Αν δεν μπορούμε να μειώσουμε το κόστος της ε, ε, γραφειοκρατίας ή της συμμόρφωσης με κανόνες ε, για εξαγωγές στην Αμερική, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και η θέση στην εξαγωγική οικονομία είναι υψηλά αμοιβόμενες, είναι ποιοτικέ και έχουν και καλύτερους μισθούς. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθούν εκεί θέσεις εργασίας ποιοτικέ με την Κορέα, όταν κάναμε την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, αυξήθηκαν οι εξαγωγέ μα τον πρώτο χρόνο κατά 15% και στου τομεί που απελευθερώθηκαν κατά 46%. Είναι ουσιαστική ευκαιρία, αν ακούσουμε τι μικρομεσαίε, να γίνει σωστά η προσπάθεια. Και χαίρομαι ε, που εστιάζει στι μικρομεσαίε η συγκήτρια. Είπαμε ότι το κεφάλαιο αυτό για τι μικρομεσαίε πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Για τις δημόσιες συμβάσεις Ίσως θα ήταν σκόπιμο και χρήσιμο να βάλουμε ε, ένα χρονοδιάγραμμα, ότι υπάρχει ανάγκη ας πούμε για την ε, αρχή προώθησης του εμπορίου για να έχουμε ένα καλύτερο, πώς να το πω, ίσως κανόνες παιχνιδιού ε, να ζητήσουμε τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Και για το θέμα της θεώρησης διαβατηρίων, α είμαστε ρεαλιστέ. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτέ εξ όσων ε, κατάλαβα, δεν μπόρεσαν να ε, το διαπραγματευτούν εκεί, αλλά υπάρχει η λύση της Αυστραλίας που είχαμε παράλληλε συζητήσει για ποσοστώσει. Αυτό μπορεί να βοηθάει με κάποιο είδους αμοιβαία αναγνώριση και για τις υπηρεσίες. Πάντως είναι ενδιαφέροντα τα σχόλια που ακούσαμε και συμφωνώ ότι θα πρέπει να εκφράσουμε και τις ανησυχίες και τις επιθυμίες μας. Θα λόγω και πάλι στην εισηγήτρια για να ακούσουμε και τα δικά της σχόλια. Ευχαριστώ. Μία γενική παρατήρηση. Η συζήτηση απέδειξε ότι το TTIP είναι σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας και ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας εδώ μέσα, ίσως με πιο δομημένο τρόπο, κεφάλαιο το κεφάλαιο και μετά από πληροφόρηση και της Κομισιόν. Γιατί μερικά ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν μόνο από την Κομισιόν, όχι από μένα. Πάντως θα λάβω σοβαρά υπόψη μου όλα σας τα ερωτήματα τώρα δύο-τρία σημεία που τέθηκαν από πολλούς. Για την προστασία των καταναλωτών. Είναι ευαίσθητο θέμα νομίζω και μπορεί να γίνει και ακρόαση για αυτό το θέμα θα γίνει ακρόαση για το θέμα με διαφορετικούς ομιλητές, διάφορους ομιλητές από διάφορες οργανώσεις καταναλωτών για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τι παίζεται. Η ορολογία που χρησιμοποιώ, η διατύπωση είναι ότι θέλουμε να προωθήσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην Ευρώπη και συμφωνώ με την Κατρίν ότι πρέπει να τα βρούμε σωστά και να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση που ταυτόχρονα να στέλνει το μήνυμα όπως είπαν και οι συντηρητικοί, ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες ως Ευρωπαίοι καταναλωτές, αλλά επίσης ότι το επίπεδο, το υψηλό επίπεδο προστασίας που έχουμε εμείς δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Για τις δημόσιες προμήθειες εξετίμησα ιδιαίτερα αυτά που είπε ο συνάδελφος Ταραμπέλα που ήταν και εισηγητής για αυτό το θέμα παλαιότερα και εξήγησε πολύ καλά πώς έχει η κατάσταση στην Ευρώπη και πώς στις Ηνωμένε Πολιτείες. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο υψηλά ενδιαφέροντα και συμφέροντα της Ευρώπης Άρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη διατύπωσή μας έτσι ώστε να φαίνεται τι σημασία δίνουμε και στο θέμα των δημόσιων προμηθειών. Τι regulatory. Για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της συνεργασίας, της ρυθμιστικής συνεργασίας. Δηλαδή, αν συμφωνήσουμε κάτι να είναι δεσμευτικό. Αν όμως δεν υπάρξει συμφωνία, παρόλα αυτά θα διατηρήσουμε την αυτονομία μας στις ρυθμίσεις μας. Και τέλος, ξέρω τώρα ότι ανοίγω το κουτί της Πανδώρας, το ISDS που είναι το πιο ευαίσθητο θέμα πολιτικά, όλοι το ξέρουμε αυτό θα πρότεινα τη συζήτηση αυτή να την αφήσουμε στην, διακομα... στην Επιτροπή Ίντα που είναι η υπεύθυνη επί της ουσίας και τη γνωμοδότησή μας στη γνωμοδότησή μας στο μήνυμά μας να βασιστούμε στα ουσιώδη θέματα που αφορούν καταναλωτές και επιχειρήσεις. Δεν λέω ότι ο ISBS δεν είναι σημαντικό και για αυτούς αλλά δεν είναι όλα τα θέματα δικής μας δικαιοδοσίας, ενώ είναι σημαντικά και για τους καταναλωτές. Νομίζω όμως ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη δομή της έκθεσης ΙΝΤΑ και να τονίσουμε ιδιαίτερα εμείς τα θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία μας. Τώρα θα ήθελα να σας καλέσω στην ακρόαση που οργανώνουμε και προσβλέπω στα σχόλιά σας και στην επόμενή μας συνάντηση με τους Σκιώδης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Φαίνεται πόσο σημαντική είναι η συζήτησή μας. Ξέρω ότι ο κύριος Χίντεχουπ από την Κομισιόν έχει έρθει να ακούσει τη συζήτηση. Μήπως θέλει να σχολιάσει και τίποτα. Ευχαριστώ. Τμήματάρχης. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε πολλές, πολλή δουλειά στην ημερήσια διαταξή σήμερα το πρωί βέβαια, αλλά πρέπει να κάνω και εγώ λίγε παρατηρήσει για να σα διευκολύνω στην εξέταση του κειμένου σα. Για μερικά επιμέρου σημεία, για τη διαφάνεια. Να επιστήσω την προσοχή σα. στα πολύ σημαντικά νέα μέτρα που έχουμε εγκρίνει τι τελευταίε 8 εβδομάδε, ώστε να διατίθενται στο διαδίκτυο όλα μα τα έγγραφα Εκεί όλες οι ευρωπαϊκές προτάσεις μπορούν να, να αναγνωστούν από όποιον θέλει και έτσι υπάρχει διαφάνεια και φαίνεται τι ακριβώς θέλουμε και στους τελικούς στόχους αλλά και το συγκεκριμένο πλαίσιο που ζητούν και οι Αμερικανοί συνομιλητέ μα. Θα τα δείτε στο διαδίκτυο και τα τεχνικά αυτά έγγραφα συνοδεύονται από fact sheets, με έγγραφα δηλαδή με τεχνικά στοιχεία. Οπότε θα σας τα συνέστηνα. Και για τα τελικά κείμενα υπάρχει πρόσβαση για τους βουλευτές του σώματός σας και για τα μέλη της Επιτροπής ΙΝΤΑ και για μέλη άλλων επιτροπών ανάλογα με το κείμενο επί το οποίο έχουν δικαιοδοσία και αρμοδιότητα οι επιτροπές. Κάποια σημεία τώρα. Ε, η ρυθμιστική συνεργασία και ο σχετικό στόχο που ενδιαφέρει τόσο πολύ την Επιτροπή σα. Πρώτα απ' όλα να τονίσω κάτι που νομίζω ότι είπαν πολλά μέλη δεν υπάρχει περίπτωση υποβάθμιση των προτύπων σε καμία περίπτωση. Είτε οι Αμερικανοί είτε εμείς δεν το επιθυμούμε. Ούτε υπάρχει θέμα απώλειας της ρυθμιστικής αυτονομίας. Αυτή είναι και μια σημαντική διαφορά για το πώς οργανώνουμε εμείς την ενιαία αγορά. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που ελπίζουμε να πετύχουμε με τις ΕΠΑ και την Συμφωνία TTIP είναι η συνεργασία μεταξύ των ανεξάρτητων ρυθμιστών. Αυτή η συνεργασία θα βασιστεί σε θελοντική βάση. Δεν μπορεί να γεφυρωθούν οι διαφορές και να συνεχίσουμε να ζούμε με αυτές, αλλά θέλουμε να περιορίσουμε το κόστος για την, με την περιττή επανάληψη προτύπων ή τουλάχιστον να πετύχουμε καλύτερα πρότυπα. Διότι μπορεί κανείς να μάθει κιόλας από τον συνομιλητή του στις ρυθμιστικές αρχές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βεβαίως και αυτό βρίσκεται στον πυρήνα του ενδιαφέροντός μας για, το, για τις δικαιωματεύσεις. Ιδίως για να διευκολύνουμε τις εμπορικές συναλλαγές των ε, μικρομεσαίων οι Βρίσκουν τρόπο να μπουν οι μια στην αγορά της άλλης. Είναι πιο δύσκολο αυτό για τους μικρούς. Ε, και για, την, για το μηχανισμό επίλυσης ε, διαφορών μεταξύ κρατών και ιδιωτικών επενδυτών. Ναι, υπάρχει όργανο επίλυσης ε, διαφορών με κυβερνήσεις για τις μικρότερες εταιρείες, αλλά αυτό ξέρουμε ότι έχει πολιτικές συνέπειες και μεγάλο κόστος. Υπάρχει λοιπόν συσχετισμός μεταξύ του ISDS και του μικρομεσαίου για τις προμήθειες. Να σας ε, τονίσω, γιατί και αυτό αφορά την καρδιά των εργασιών σας, ότι είναι ένας πρωταρχικός μας στόχος της διαφαματεύσης με τις ΗΠΑ. Η Ευρωπαίοι ε, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς να συμμετέχουν σε ίση βάση με τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους. Ε, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο αυτό βέβαια στην πράξη, αλλά είναι πολύ μεγάλο και το διακύβευμα. Και τέλος, εάν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο και για τον ίδιο το μηχανισμό επίλυσης διαφορών, να σημειώνω με προσοχή όσα επισηγήτρια ότι εδώ υπάρχει και αρμοδιότητα άλλης επιτροπής, αλλά όλοι σας ως βουλευτές έχετε απόψεις για το θέμα, το πρόσεξα τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε σας συστήνω θερμά την έκθεση που συντάξαμε εμείς για τον εντοπισμό των που θα μας απασχολήσουν σε μελλοντικέ εργασίες μας και στις μελλοντικές μας συζητήσεις με το Κοινοβούλιο, για να δούμε πώς θα ε, σχεδιάσουμε το ε, θέμα του μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτών, ιδιωτών επενδυτών. Δεν είναι διπολικό το θέμα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ένα ναι ή με ένα όχι. Πρέπει να κάνουμε κάτι ανάλογα με τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά και να, ε, να προβλέψουμε περαιτέρω μέτρα ε, για να ενισχύσουμε το μηχανισμό αυτό με όσα προέκυψαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές Ιανουαρίου. Εάν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, νομίζω έχουμε μια πλούσια βάση συζήτηση για να αποφασίσουμε πώς θα εξισορροπήσουμε τα διαφορετικά στοιχεία που ευσταθούν και είναι λογικό να υπάρχουν εδώ διαφορετικές απόψεις, το παραδεχόμαστε, αλλά προσπαθούμε να καλύψουμε την ουσία του θέματος, ώστε να έχουμε μια συζήτηση τεκμηριωμένη τις επόμενες εβδομάδες. και να καταλήξουμε σε μια κοινή άποψη των, ε, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επιμέρους κρατών ε, που να είναι ευρέως πεπισμένοι για το πώς θα προωθήσουμε αυτό το μηχανισμό ISDS. Δεν είναι μόνο θέμα της συμφωνίας TTIP, είναι και των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όπως προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε πρέπει να προσέξουμε πώς θα οργανώσουμε τις εργασίες με το θέμα αυτό. Και αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια θέση πολύ ιδιαίτερη, καθώς διαφορετικές απόψεις υπάρχουν από όλες τις Ευχαριστώ. Um, Εγώ ευχαριστώ πολύ και όπως είπατε ε, μας ξέφυγε λίγο το χρονοδιάγραμμα αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η γνωμοδότηση της λύσης για κοσάρι για λύσεις διαλειτουργικότητας για δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη, εταιρείε και πολίτες. Ε, είναι παρουσίαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής της πρότασής Sorry, I should have reminded you, by the way. Ήθε, έπρεπε να σας είχα πει ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι, μια στιγμή να το βρω για το TTIP, την γνωμοδότηση κυρίας Σαρανσόβα, 25 Φεβρουαρίου. Ναι, 25 Φεβρουαρίου. Συμφωνώ με τα όσα είπατε για το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Are we ready? Είστε έτοιμοι? Okay, with apologies, we've just been playing musical chairs in the committee this morning. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση και λίγο την ασάφεια που επικρατεί εδώ. Λύσεις λοιπόν διατουργικότητας για τι ευρωπαϊκέ δημόσιες διοικήσει. Ε, η αρμόδια επί τη ουσία είναι η Επιτροπή Ήτρε. Εμεί γνωμοδοτούμε, είμαστε συνδεδεμένοι βάσει του άρθρου 54 του κανονισμού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την έκθεσή τη. Καλώς ορίσατε κυρία Έγκεστάτ, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώς μας ήρθατε. Και ε, έχετε στη διάθεσή σας στο e-meeting επιγραμμικά τα στοιχεία PowerPoint της ε, παρουσίασης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, και κύριοι βουλευτές, με μεγάλη χαρά ήρθα να σας παρουσιάσω το ΆΙΣΑ. Λέγομαι είμαι διευθύντρια αρμόδια για αυτά τα θέματα στη Γενική Διεύθυνση Digit. Τι εστί λοιπόν διαλειτουργικότητα, περί τίνος πρόκειται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ορίζει ως εξής το 2010 στην ανακοίνωσή της ε, τη σχετική. Είναι βασικά πώς μπορούμε να κάνουμε δύο διαφορετικές ενότητες και μονάδες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες ουσιαστικές. Είναι πολύ απλό. Περί πρόκειται για μας καθημερινά να έχουν οι δημόσιες διοικήσεις κάποιες βασικές αρχές οι ίδιες που να τις ε, ακολουθούν. Εδώ αριστερά τις βλέπετε. Ποιες είναι αυτές οι αρχές. Να δίνονται μία φορά τα στοιχεία, ε, είναι ενιαία η θηρίδα, ε, ο σύνδεσμος ας πούμε επαφής να είναι ηλεκτρονικές υπηρεσίες κατά κανόνα και ε, να μπορούν να διασυνδέονται πολλές δημόσιες διοικήσεις για να παρακολουθούν ε, ας πούμε μια εταιρεία ή ένα πολίτη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής και να μπορούν να τον ακολουθούν. Αν τα κάνουμε όλα αυτά θα έχουμε πολύ μεγάλη διασύνδεση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, θα αυξήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και ε, περισσότερες ομάδες θα έχουν τα στοιχεία αυτά, θα τα μοιράζονται και θα χειρίζονται. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Βελτιώνεται η λήψη των αποφάσεων γιατί έχει περισσότερα στοιχεία, έχουν περισσότερες δυνατότητες και υπηρεσίες. And last οι δημόσιε διοικήσει παίζουν σημαντικό ρόλο, όπω ξέρετε, για την οικονομία και τελευταίο, χωρί αυτό να είναι το λιγότερο σημαντικό, είναι καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και έχουν περισσότερε προσβάσει στα δημόσια στοιχεία. Η διαλειτουργικότητα έχει αναγνωριστεί από το 1995 ε, ως προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, ιδρύθηκε το πρώτο πρόγραμμα, το AIDA. Τώρα είμαστε τόσα χρόνια μετά και βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Γι' αυτό μας ενθαρρύνει να προταθεί το ΆΙΤΑ στο τετράγωνο ως διάδοχο πρόγραμμα ε, για να δούμε τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο πεδίο αυτό στην Ευρώπη. Η ΆΙΖΑ ε, στο τετράγωνο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014. Ποιο είναι το πρόγραμμα και τι κάνει. Έχει ένα στόχο ενιαίο όπως και το προκάτοχο πρόγραμμα λύσεις διαλειτουργικές που υποστηρίζουν την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών της Ευρώπης που είναι οι άμεση δικαιούχοι αλλά και μεταξύ και ε, της διοίκηση και των πολιτών οι οποίοι πλέον πολίτες είναι οι έμεση δικαιούχοι και αυτή είναι η καινοτομία θέλετε και η ρητή αναφορά στους πολίτες. Ε, το πεδίο εφαρμογής διευρύνεται και όπως το προκάτοχο πρόγραμμα ε, θα εντοπιστούν, δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν λύσεις διαλειτουργικότητας απεριόριστης χρήσης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν την υλοποίηση και εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης θα διευρύνει τις δραστηριότητες αυτές και θα τις εδραιώσει. Ταυτόχρονα θα είναι και ένας εποαστήρας, ένας ολαπτήρας λύσεων για να οριμάζουν και να μπορούν να εφαρμόζονται από τους διάφορους διάβλους παροχής υπηρεσιών. Και επίση να μπορούν αυτά τα συστήματα ε, να πηγαίνουν σε άλλα που ισχύουν όπως το ΣΕΦ και να γίνεται αυτό το migration. Έχουμε λοιπόν ενιαία προσέγγιση έχει και λειτουργικούς στόχους με προγραμματικές δράσεις δηλαδή. να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν λύσεις που ήδη λειτουργούν και υπάρχουν όπως το πρώτο ΆΙΖΑ. Επίσης, επαναχρησιμοποίηση νέων διατομεακών ή διασυνοριακών λύσεων όπως επίσης ισχύει και στο ΆΙΖΑ. Εκτίμηση των επιπτώσεων όταν εγκρίνεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως και στο παλιό Άιζα. Αλλά ποιο είναι το νέο τώρα να εντοπίσουμε νομοθετικά κενά που εμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δημοσίων ε, διοικήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έιρα ε, είναι το θέμα της αρχιτεκτονικής αναφοράς και η iCard που είναι μια χαρτογράφηση λύσεων που μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν εγκριθεί και εφαρμοστεί. Επίσης, ε, το θέμα των κοινών προδιαγραφών και προτύπων είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του ΆΙΖΑ στο τετράγωνο και ε, να δούμε μηχανισμούς που θα μετράνε και θα ποσοτικοποιούν ε, τα ωφέλη, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι είναι υποφελείς οι λύσεις που υιοθετούνται. Ε, το πρόγραμμα επίσης θα υφίσταται συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση και μάλιστα επιγραμμικά είναι πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Θα υπάρχει μια ενδιάμεση αλλά και μια τελική ε, αναθεώρηση, ε, αποτίμηση μάλλον που θα σας υποβληθεί. Και στην νομοθετική πρόταση έχουμε προβλέψει και δείκτες για να μετράμε το πρόγραμμα και τι αποδίδει και θα, ποιοι είναι οι βασικοί διευκολυντές, enablers. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ λειτουργικό, είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ποσοτικά λοιπόν μας ενδιαφέρει να μετράμε ποιο είναι το όφελος για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Βλέπετε τον προπολογισμό εδώ για την εφαρμογή, είναι πενταετές το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος MFF 131 εκατομμύρια ευρώ είναι ε, το ποσό που έχει εκεί δοθεί. Ετησίως κατά μέσο όρο 26 εκατομμύρια όπως και το παλιό πρόγραμμα ΆΙΖΑ για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των μέτρων που ήδη έχουν υιοθετηθεί. Για να δούμε και το πολιτικό πλαίσιο τώρα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι το δημόσιο, ο δημόσιο τομέα είναι βασικός παράγον στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και, ε, και είναι και τμήμα της λύσης αυτό για την οικονομική κρίση. Το μισό ΕΠ στην Ευρώπη ε, δημιουργείται από το δημόσιο τομέα. 25% της νεολικής απασχόλησης είναι εκεί και 19% του ΕΠ της Ένωσης είναι οι δημόσιες συμβάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και τεράστια ποσά καταλαβαίνετε σημαίνει για τα κράτη-μέλη. Ε, ποια είναι η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα στις δημόσιες διοικήσεις. Δεν είναι και τόσο τεράστια. Αλλά υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είτε άμεσα είτε έμεσα επηρεάζουν ε, το δημόσιο τομέα και αυτό είναι η στρατηγική 2020, η ψηφιακή η αγορά, η ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και η ετήσια ε, έκθεση για την ανάπτυξη το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ο εξυγχρονισμός των Ευρωπαϊκών Δημοσίων Διοικήσεων. Δηλαδή, υπάρχουν πολιτικά κίνητρα και ενδιαφέρον για να συνεχίσει αυτή η διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη. Εδώ δεν βλέπετε τις λεπτομέρειες αυτή τη διαφάνεια, αλλά είναι μια μελέτη που δείχνει πόσος χρόνος θα εξοικονομηθεί από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις και αυτό μεταφράζεται σε οικονομίες του ΑΕΠ και με βάση πίνακες της Παγκόσμιας Τράπεζας. Είναι πραγματικά εύγλωτα τα παραδείγματα. Κοιτάξτε το Βέλγιο. Αν υπάρξει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στις δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να εξοικονομήσει 2,35 δισεκατομμύρια εκατομμύρια, η Γαλλία 12,8. Είναι πολλά τα λεφτά. Τεράστια ποσά. Και μόνο παραδείγματα για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Αν είναι λοιπόν τόσο σαφή τα ευεργετήματα, γιατί δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Ποια είναι τα εμπόδια και τι πρέπει να γίνει. Υπάρχει δεδομένη η πολιτική βούληση, ε, υπάρχει η τεχνογνωσία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σουηδία είναι από τις υψηλότερες χώρες σε διαδικτύου και χρήση. 93% των οικοκυριών έχουν ίντερνετ στη Σουηδία. 72% του πληθυσμού το χρησιμοποιούν για να συναλλάσσονται με τις δημόσιες αρχές. Αλλά όταν πρόκειται για την συνεργασία, την επιστροφή από τις δημόσιες διοικήσεις, ας πούμε μια φορολογική δήλωση που έχει συμπληρώσει online ο καταναλωτής, ο πολίτης, είναι μόλις 46%. Δηλαδή ε, υπάρχουν τα προσυμπληρωμένα έντυπα που υποβάλλουν οι πολίτες, αλλά από εκεί και πέρα η ανταπόκριση της διοίκησης ε, δεν είναι η επιθυμητή. Έχουμε περάσει στην ψηφιακή εποχή αλλά ε, είναι ad hoc κάθε φορά οι ψηφιακές λύσεις και είναι δύσκολο ε, να εφαρμοστούν από τις διάφορες δημόσιες αρχές που είναι 400 παρακαλώ τον αριθμό στην Ευρώπη. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν λύσεις που από την αρχή να είναι διαλειτουργικές. Ανεξαρτήτως της υποδομής θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική, ολιστική, όπως λέγεται, καθολική προσέγγιση. Επίσης θελήσαμε να σας δείξουμε αυτή τη διαφάνεια, τρεις διαφορετικές λύσεις. Θα τις θυμάστε όλοι, τις αναγνωρίζετε τόσο σημαντικέ Η Ευρώπη σας, Your Europe, It και IMI. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τα βλέπετε. Ε, είναι όλο και πιο επιτυχημένα μέσα και εργαλεία διαλειτουργικότητας, διασυνοριακής και όλα αυτά τα υποστηρίζει το ΆΙΖΑ. So, final uh, ε, και ε, το συμπέρασμα. Η διαλειτουργικότητα είναι κομβική για να δημιουργηθεί στρατηγική στις δημόσιες διοικήσεις, βάζει ένα πλαίσιο για να μπορούν να οικοδομούνται οι διοικήσεις και να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν η διαλειτουργικότητα δεν είναι μόνο πληροφορική, έχει να κάνει και με τις πολιτικές αποφάσεις και την οργανωτική δομή της κάθε διοίκησης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα δεδομένα. Για να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα χρειάζεται μεταρρύθμιση, αναδιάρθρωση των διοικήσεων και των μεθόδων και αυτό απαιτεί σαφείς πολιτικές αποφάσεις και βούληση για να υπάρχει μια πραγματική ενιαία αγορά για να λαμβάνεται υπόψη η διαλειτουργικότητα από την αρχή, από το σχεδιασμό των ναι, ναι, ναι. υπηρεσιών και ε, των λύσεων. Και εκεί μπορεί να βοηθήσει το ΆΙΖΑ στο τετράγωνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας που την έχουμε και εμείς ψηφιακά, ψηφιακά στην ιστοσελίδα μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέγει η Μιλήτρια, για την σαφέστατη παρουσίασή της. Κομισιόν, Τα θέματα αυτά είναι τεράστια προτεραιότητα φαίνεται της Κομισιόν και ορισμένων χωρών μελών. Οι εξελίξεις κινούνται ταχαίως και ορισμένοι το βρίσκουν δύσκολο να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει στην κατακερματισμένη, στο κατακερματισμένο ευρωπαϊκό ψηφιακό πρόγραμμα. Στο δε των επιτρόπων υπάρχει και εκεί σύγχυση και υπερκάλυψη, αλλά πρέπει να υπάρξει επιτέλους κάποιος κεντρικός συντονισμός. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή ΕΜΚΟ είναι ιδεώδες εργαλείο για να γίνει αυτός ο συντονισμός, ο συντονιστικός ρόλος για να διασφαλιστεί ότι το θέμα δεν θα θεωρηθεί καθαρά τεχνικό. Κρίμα που έγινε τέτοια καθυστέρηση και πόλεμος μεταξύ Ήτρα και Ήμκο. Γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα η Ήτρα και η Ήμκο συμμερίζονται δικαιοδοσίες και αυτή είναι και η σωστότερη λύση. Το ίσο 2 είναι, έχει τεχνικό χαρακτήρα αλλά δεν είναι αυτό λόγος για, να, για απογοήτευση ή απεσιοδοξία. Πρέπει να δούμε τις δυνατότητες που έχει η ενιαία αγορά. Συμφωνώ με την Κομισιόν εγώ. Κομισιόν. Ότι δεν μπορούμε να αποτύχουμε, δεν έχουμε τα μέσα να αποτύχουμε. Χάσαμε πολύ χρόνο και προσπάθειες και εντεύρα για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Χαιρετίζω το ότι το ότι λέγω το ίσο 2 έχει επεκταθεί για να καλύπτει χρήστες και ακόμη και η λέξη πολίτης αναφέρεται εδώ, πολίτης. Mm. Είναι καλύτερο αυτό, αυτή η φευγαλαία αναφορά είναι καλύτερη από το τίποτα. Και βεβαίως τελικά όλα αφορούν τους πολίτες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η προοπτική των πολιτών πρέπει να έρχεται στο προσκήνιο πιο συχνά. Έχουμε τρομερή πίεση χρόνου. Πρέπει να καταλήξουν όλα αυτά σύντομα. σύντομα. Το ίσο 1 λίγησε λίγο. Και φυσικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρήσουμε το αυστηρό αυτό χρονοδιάγραμμα. Αλλά πρέπει η Κομισιό να ξέρει ότι πρέπει να σέβεται τα σαρχάς της δημοκρατίας και να μην προσπαθήσει να μας το περάσει σαν οδοστρωτήρα. Χρειαζόμαστε χρόνο για να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Αλλά βέβαια φταίμε και εμείς και εμείς. Διότι αυτοί οι πόλεμοι μεταξύ επιτροπών μας καθυστέρησαν πολύ. Έχω λοιπόν τα ερωτήματά μου. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τη βασική ιδέα. Βασική ιδέα. Ποια είναι τα όρια της πρότασης της Κομισιόν. Είναι κάτι καθαρά τεχνικό. Είναι τρόπος κατανομής πόρων για συγκεκριμένα προγράμματα ή μήπως, μήπως εσείς στην Κομισιόν το θεωρείτε σαν κάτι βαθύτερο, σαν κάτι που θα έχει περισσότερες επιπτώσεις από ό,τι φαίνονται. Μήπως θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι ως προς την πιθανή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών και δημοσίου τομέα. Μήπως και μήπως επίσης θα μπορούσατε να μας πείτε μερικά περισσότερα πράγματα για το πώς σκοπεύει η Κομισιόν να μοιράσει αυτούς τους πόρους. Με τι κριτήρια. Τι. Και αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα για το TTIP και για αυτό το θέμα είναι το εξής Συνεχώς επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα. Γιατί τα ανάλαβε όλα αυτά η Γενική Διεύθυνση ΨΥΦ, digit, διότι θέλουμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την διάδραση μεταξύ αυτή, τη σύνδεση μεταξύ αυτού του προγράμματος και του Connecting Europe ας πούμε. Europe. και ποιος θα έχει τη γενική ευθύνη. Και αυτό είναι σημαντικό ερώτημα. Σας κατευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και τώρα για το ΕΛΚ η κυρία Πάουνοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξωτική παρουσίαση και επίσης την, την εισηγήτρια την κυρία Κουνσάρη για τα σχόλιά της. Ήδη έχουμε αρχίσει τη συνεργασία με τις υπηρεσίε τη και με την ομάδα των συνεργατών της και την ίδια να μένουμε να συνεργαστούμε με ανυπομονησία. Καθώ και με τις πιο γιατί μας ε, μπώνει στην Επιτροπή Ήτρε. Χθε το ΕΛΚ οργάνωσε μια κρόση για την ενιαία αγορά. Ακούσαμε εκεί ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα των κυβερνήσεων είναι πολύ σημαντικά για την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς και η Επίτροπος Μπιενκόφσκα είπε ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι από τα σημεία κλειδιά για το σκοπό αυτό. Θα επικεντρωθώ σε τέσσερα σημεία. Το πρώτο θα ήταν μάλλον πώς να μεταδώσουμε τα ωφέλη των προγραμμα... του προγράμματος στους συμπολίτε μας. Υπάρχουν θετικά παραδείγματα όπως στη Σουηδία που αναφέρθηκε, αλλά και στη Σουηδία ακόμα που έχει τη μεγαλύτερη δίσδυση από διαδίκτυο από τις δημόσιες υπηρεσίες ε, έχουμε μόνο 46% παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πώς λοιπόν να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων για περισσότερες ηλεκτρονικές λύσεις. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ε, από την πολιτική σκοπιά επίσης του ΆΙΖΑ Πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί σωστά και είναι αποφελές για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι όταν λειτουργήσει σωστά το σύστημα του e-government τη ηλεκτρονικής κυβέρνηση, οι πολίτες μπορεί να ωφεληθούν, αλλά πόσο το γνωρίζουν είναι το άλλο ερώτημα. Νομίζω ότι το προτινόμενο χαρτοφυλάκι για την υλοποίηση του προγράμματος ΆΙΖΑ 2 για την περίοδο 2016-2020 131 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω λοιπόν ότι αν έτσι είναι, τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μεταδώσει καλύτερα στους πολίτες τα ωφέλη του προγράμματος αυτού. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης ο στόχος της επικοινωνιακής στρατηγικής υπάρχει. Πώς θα μεταφραστεί αυτό το τεχνικό καταπτυσμένο κείμενο σε κάτι πιο εύληπτο για τους πολίτες. Επίσης, κάποια από τα μέλη που βρίσκονται εδώ ίσως έπρεπε να προβλέψουν συναντήσεις με τους εκλογείς τους, τις εκλογικές της περιφέρειες, που ε, καλό θα ήταν να γνωρίζουν τα θέματα του προγράμματος αυτού. Μόνο εάν έχουμε συγκεκριμένα από τα παραδείγματα θα πείσουμε για τα ωφέλη του προγράμματος. Επίσης να σταθώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι κάτι που μας λείπει στο κείμενο της πρότασης, αν και προστέθηκε στον τίτλο του εγγράφου, ώστε να ωφελήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα όμως να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις μικρομεσαίες. Και επίσης μεγαλύτερη προσοχή θα έπρεπε να δοθεί στην επαναχρησιμοποίηση των δημοσίων δεδομένων που θα ε, ε, αξιοποιούνται από πολίτες και επιχειρήσεις. Καθώς οι μικρομεσαίες είναι ένας βασικός παράγοντας της αγοράς που έχουν πληγεί περισσότερο από τα οικονομικά βάρη, άχθη, θα πρέπει να έχουμε υπόψη όταν σχεδιάζουμε λύσεις και αξιολογούμε το πρόγραμμα και τις δικές τους ανάγκες. Να μην μιλούμε για τις επιχειρήσεις ε, γενικόλογα, αλλά πιο συγκεκριμένα. Επίσης, είμαι υπέρ μιας αιτήσεως αναθεώρησης της υλοποίησης του προγράμματος ΆΙΖΑ 2 και όχι μόνο από την Επιτροπή ΆΙΖΑ, ΆΙΖΑ 2, αλλά και από το Ευρωκοινοβούλιο. Και τελευταία μου παρατήρηση για την ουδετερότητα του δικτύου. Αυτό είναι άλλο ένα θέμα που θα πρέπει να σκύψουμε με προσοχή. Στο κείμενο καθώς το διαδίκτυο και η τεχνολογική ιδιωτερότητα είναι σημαντικότατα. Λίγο πολύ αυτές ήταν παρατηρήσεις μου ως αυτή τη χρονική στιγμή. Είμαι θετικά διακείμενη προς την ολοκλήρωση εξέτασης του προγράμματος και την υλοποίησή του στο τέλος του 2015 να μην χάσουμε όσα έχει πετύχει ως τώρα το ΆΙΖΑ 1. Ευχαριστώ. Thank you and I've been... Ευχαριστώ. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για το θέμα, για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές και νομίζω ότι θα ήταν καλό να θυμίσουμε σε όλους γιατί το εξετάζουμε αυτό. Το εξετάζουμε γιατί θέλουμε τις καλύτερες δυνατές δημόσιες υπηρεσίες που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικονομίας του 21ου αιώνα. Να λειτουργεί το ψηφιακό στοιχείο εξορισμού ε, για τους πολίτες στην Ευρώπη και να γνωρίζουν ότι έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες αυτή και ότι είναι και ασφαλής και προστατευμένοι. Αυτό είναι ο στόχος της διαλειτουργικότητας. Είναι ένα μέσο για να καταλήξουμε στο σκοπό, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός. Ο αυτός σκοπός είναι να έχουμε την βέλτιστη προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό θέλουμε μια ψηφιακή ε, μεταμόρφωση σε όλη την Ευρώπη για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτή η μεταμόρφωση δημιουργεί απαιτήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο. Όλοι οι δημόσιοι φορεί, οι περισσότεροι μάλλον, χρησιμοποιούν το εθνικό επίπεδο, το αξιοποιούν και επιτρέπουν στους πολίτες να επικοινωνήσουν και να έρθουν σε διάλογο με το σύστημα σε μια πρώτη φάση, ενώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε μόνο ένα, μια συνιστόσα όλου αυτού του συστήματος, αλλά είναι μόνο τμηματικό αυτό. Θέλουμε λοιπόν να θυμηθούμε όλοι ποιος είναι ο τελικός στόχος εδώ. Ε, πέραν αυτού είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερα, ε, να βασιστούμε περισσότερο στις ανάγκες, στη ζήτηση δηλαδή που εκφράζεται, και να δώσουμε έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε άλλους τελικούς χρήστες. Δηλαδή ε, να κατευθύνει το σχεδιασμό μας η ζήτηση, οι ανάγκες, όχι μόνο ορισμένε ε, λιγάριθμες ε, στοχευμένες υπηρεσίες. Να είμαστε σίγουροι ότι δημιουργούμε μια τέτοια πλατφόρμα που μπορεί να έχει μεγαλύτερε διαστάσει αν χρειαστεί, να μην είναι περιορισμένη με αυτά υπόψη να μας οδηγήσει η διάσταση της ζήτησης και να είμαστε πιο στοχευμένοι. Βρίσκω ότι είναι κρίμα που δεν υπήρξε η μελέτη αντικτύπου και διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους πριν τη στιγμή που θα υποβαλόταν η πρόταση. Ε, εντάξει θα μου πείτε είναι το ΆΙΖΑ 2, δεν είναι το ΆΙΖΑ 1, δεν είναι νέα πρόταση, <laughs> είναι μια συνέχεια προηγούμενης, ε, προηγούμενου προγράμματος, όμως και πάλι πιστεύω ότι θα είχαμε ωφεληθεί Εάν είχε γίνει μια ενδελεχής αποτίμηση τη προηγούμενη φάση. μιλάμε για το χρήμα των φορολογουμένων, μιλάμε για δημόσιε υπηρεσίε σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό πολλέ φορέ πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο διάλογο εκεί είναι άριστος. Δηλαδή τα ωφέλη προκύπτουν όταν αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό μας. Αυτές είναι οι αρχικές μου παρατηρήσεις και καλωσορίζω και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων σε σχέση με την πρόταση. Σας προσκαλώ. Ρότζερ. Ευχαριστώ κύριε Γιακοντσάρη. Και προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους κοιόδης. Το σημαντικότερο είναι να κατανεμηθεί η πληροφόρηση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Έχω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Πώς βελτίωσε το ΆΙΣΟ το άισα την ε, εποπτεία των αγορών. Στα. Α, σύντομος και καλός. Είναι κανείς άλλος εδώ για να μιλήσει έτοιμος. Πρόθυμος η κυρία Κάλλας. Και εγώ νομίζω ότι το ISA είναι σημαντικό πρόγραμμα για να βελτιωθεί η διοίκηση πανενωσιακός Και είναι σημαντικό να γεφυρώσουμε με διαφορετικούς μεταξύ τους στόχους, όπως την τα προμήθειες. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάπτυξη ή τα λύσεων για πιο αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και για να είναι πιο ασφαλή τα συστήματα. Όπως είπε και η Εύα προηγουμένως, πρέπει οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη όμως στο σύστημα. Να μην ανησυχούν μήπως τα δεδομένα τους online δεν είναι ή ασφαλέστερα από ό,τι στο χαρτί. Επομένως πρέπει το ISA να παίξει ένα ρόλο οθώντας τα κράτη-μέλη να βρουν λύσεις για να προστατεύονται τα δεδαμένα των πολιτών. Uh, so, ε, Ας πούμε να υπάρχει ένα σύστημα πιστοποίησης ε, που να είναι ασφαλές. Επίσης το θέμα του πώς θα το πουλήσουμε αυτό στο κοινό, πώς θα πείσουμε το κοινό να έχει ο πολίτης μία μονοαπευθυντική θηρίδα που λέμε για, να, για τα θέματα αυτά. Και τέλος, είναι επίσης σημαντικό να μην αρχίσουν από το μηδέν όλες οι Ιταλίσεις Παραδείγματος χάρη στην Εσθονία το ασφαλές σύστημα που δημιουργήσαμε για τις ΙΤΑ πληρωμές χρησιμοποιήθηκε σε όλη μας τη διοίκηση όσον αφορούσε την Ένωση. Και η εμπιστοσύνη είναι το κυριότερο στοιχείο για την χρήση των υπηρεσιών αυτών από τους πολίτες. Πρέπει όμως να είναι και βολικές και να έχουν την εμπιστοσύνη ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές των υπηρεσίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει να επανέλθει σε τίποτα. Ζητή, ζήτη, ζήτη. Ζήτρια, ζήτρια. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Πάρα πολύ χρήσιμα φυσικά για μας, πολύτιμα. Θα επανέλθω για ένα συγκεκριμένο, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ε, ήθελα, μου επιτρέπετε, να αρχίσω από τα όσα είπε η συγκήτρια για τον κατακαιρματισμό των αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι χρειάζεται ένα κεντρικό σημείο συντονισμού και η Επιτροπή σας θα ήταν ε, κατάλληλη. Το ίδιο κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εγκάρσια προσπάθεια μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καμιά φορά είναι δύσκολο να διακριθούν οι αρμοδιότητες και να συντονιστούμε για να έχουμε αποτέλεσμα. Υπάρχει μια ευκαιρία λοιπόν τώρα με το ΆΙΣΑ 2 ε, Χρειάζεται μια ομάδα συντονισμού όντως, αλλά δεν έχει ακόμα συσταθεί για να καλύπτει όλα τα διάφορα σημεία του εξχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και του δημοσίου τομέα γέννη. Το προωθούμε και το παρακολουθούμε καθημερινά. Θα βοηθήσει και αυτό. Θέλω να το τονίσω γιατί έχει σημασία και για τη μεταξύ μας συνεργασία. Γιατί η διάδραση ΆΙΖΑ και διευκόλυνση ε, Connecting Europe. Ε, το ΆΙΖΑ είναι η προετοιμασία ακριβώς για το ΣΕΦ. Δεν επικαλύπτονται, αλλά διασυνδέονται ε, χωρίς ε, καμία δυσαρμονία. Το ISA δημιουργεί κάποιες μονάδες, building blocks, για να ε, προχωρήσει μετά ε, στο ΣΕΦ. Και επίσης εργάζεται σε ένα πλαίσιο προτύπων. Είναι διπλή η δράση του ISA. Είμαστε και με το ΣΕΦ, το επιχειρησιακό τμήμα, σε συνεργασία που είναι και αυτό στη Γενική Διεύθυνση Digit ε, ε, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε στενή επαφή με όλες αυτές τις προσπάθειες. Για την ψηφιακή ενιαία αγορά τώρα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό η διαλειτουργικότητα. Ε, ε περιέχεται σε, στις περισσότερες θα έλεγα από τις δράσεις που προτείνουμε. Είναι πάνω μια υποκείμενη προσπάθεια. για τη μελέτη αντικτύπου. Ισχύει ότι δεν έχει γίνει επειδή είναι συνέχιση προηγούμενου προγράμματος. Το ΆΙΖΑ τώρα είναι ΆΙΖΑ στο τετράγωνο, το δεύτερο. Και την εξάντε evaluation των εκ των προτέρων ας πούμε έλεγχο κάναμε για να δούμε τι θα μπει στο δεύτερο πρόγραμμα. Είχαμε πολλούς γύρους διαβουλεύσεων ατύπων όσο και επισήμων για να δούμε ποιο θα είναι το περιεχόμενο του νέου προγράμματος. Πολλή δουλειά έχει γίνει, πιστέψτε με, ακόμα και αν αυτό δεν είναι ε, με τυπική μελέτη αντικτύπου. Η μελέτη αντικτύπου χρησιμοποιείται για να εντοπιστεί ένα πρόβλημα και να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση. Εμείς εδώ επιλέξαμε ένα άλλο τρόπο αξιολόγησης και αποτίμησης για να δούμε πώς, ε, τι συνέχεια θα δοθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα. κάναμε και μια ενδιάμεση αναθεώρηση του πρώτου Άιζα ε, και αυτό μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσουμε στο δεύτερο. Για την ασφάλεια. Γιατί το αναφέρατε ή το υπενηχθήκατε πολλές φορές. Ε, το πρόγραμμα ΆΙΖΑ, αυτό καθ' αυτό, σέβεται το κανονισμό 45 του 2001 η διαχείρισή του και η καθημερινή λειτουργία του. Υπάρχουν μελέτες, ε, κατευθυντήριες γραμμές, λογισμικό κτλ. που σέβονται πάντα την προστασία των προσωπικών δεδομένων από την αρχή. Δηλαδή από το ίδιο το σχεδιασμό το πρόγραμμα αυτό προστατεύει την ιδιωτική ζωή και εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων. Και οι δημόσιες αρχές που το χρησιμοποιούν θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι σε όλες τις εφαρμογές προστατεύεται η ασφάλεια. Από την αρχή και πάλι, από χέρι, για να λειτουργήσει με τον σωστό τρόπο. Την υλοποίηση την έχουν στα χέρια τους, καταλαβαίνετε, τα κράτη-μέλη που επιλέγουν την εκάστοτε λύση. Θα εκδώσουμε όμως κατευθυντήριες γραμμές για να ε, δούμε και αυτά τα θέματα της ασφάλειας. Θα ήθελα τώρα να αφήσω να συνεχίσει ο συνάδελφός μου για τα θέματα επικοινωνίας. σε ό,τι αφορά την επικοινωνία να σας πούμε ότι υπάρχει σχετική δραστηριότητα στο τρέχον πρόγραμμα για να ενημερώνουμε για τα πλέον του προγράμματος του πολίτες, της δημόσιας και των επιχειρήσεις. Αυτό θα ισχύσει και για το ΆΙΖΑ 2. Δεν είναι μεγάλο μέρος του προπολογισμού που προβλέπεται. Ένα εκατομμύριο ετησίως προβλέπεται για την επικοινωνία και αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα εδώ, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Όλα τα θέματα που θα θέλαμε να μεταδώσουμε, διότι μιλάμε για διαλειτουργικότητα, μια έννοια που δεν μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή από τους τελικούς χρήστες και λύσεις που επηρεάζουν την ε, μέση φάση προσφοράς των υπηρεσιών και όχι την τελική που αφορά πιο πολύ τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό έχουμε ετοιμάσει κάποια πολύ απλά βιντεάκια για να μεταδοθούν όλα αυτά με απλά λόγια και να δείξουμε στους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι τους δίνουμε προσοχή. Έχουμε μια σειρά από βιντεάκια που θα αποσταλούν σε όλες τις δημοσιοστικήσεις και θα μεταδοθούν και από τα τοπικά μέσα ενημέρωση των κρατών μελών για να υπάρξει σχετική ευαισθητοποίηση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για τους συναδέλφους που μόλις ήρθαν. Έχουμε ένα μεσάωρο καθυστέρηση γιατί είχαμε μια πολύ πλήρη συζήτηση για το θέμα του TTIP, το θεωρήσαμε σημαντικό. Υπήρχαν πολλές παρεμβάσεις. Ε, κύριε θέλετε να σχολιάσετε για το προσπαθήσω να προλάβω την καθυστέρηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για την επικοινωνία πάνω απ' όλα. Θα ήθελα να πω ότι ε, για την ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, υπάρχουν πολύ μεγάλες και πανάκριβες δημοσιεύσεις σε εφημερίδες. Ε, ήταν πολύ δύσκολο για τους πολίτες να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Βγάλανε πολλά λεφτά κάποιες διαφημιστικές εταιρείες. Ελπίζω ε, ο, ο πολίτης να αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Το είπαν και οι σκιώδεις ε, οι Είναι πολύ δύσκολο ο κόσμος, οι πολίτες να καταλάβουν τι γίνεται και πώς η δημόσια διοίκηση θα βελτιωθεί με την ψηφιακή αυτή μορφή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό είναι να κάνει μελέτες, αλλά ξέρουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν αναλφάβητοι. Και θα σας εκπλήξει ο αριθμός ε, των ανθρώπων που δεν ξέρουν καν να διαβάζουν, πόσο μάλλον χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα. Δεν έχουν ούτε υπολογιστή. Ναι, ναι, δεν ναι. Ε, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες ας πούμε, φορολογική δήλωση, κάποια συναλλαγή με νοσοκομεία ή έγγραφη στο σχολείο, αν όλα αυτά γίνουν ψηφιακά, θα ε, παραγωνιστούν ε, πολλοί πολίτες και θα βρεθούν στο περιθώριο. Θα πρέπει να γίνει έρευνα και γι' αυτό, πώς είναι οι αναλφάβητοι και πώς είναι οι ψηφιακά αποκλεισμένοι. Η κυρία Κάλας είπε δύο λόγια για την προστασία των δεδομένων. Στο Κοινοβούλιο είναι ένα θέμα αυτό που άπτε τη αρμοδιότητα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, ελευθεριών και όχι της δικής μας. Ε, και σίγουρα θα ασχοληθεί με αυτό. Την άλλη εβδομάδα στο Στρασβούργο, στις 11 του μηνός συγκεκριμένα, θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με τους σκιώδεις ηγητές για αυτό το θέμα. Με το σχέδιο της έκθεσης δηλαδή. Και κανονικά μέχρι τις 3 Μαρτίου θα έχουμε τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέρουσα συζήτηση. Thank you. Um... Ευχαριστούμε. Επόμενο σημείο στην εμπειρία διάταξη. Αντώνιο Λόπες Ιστούρι Βάιτ. Έκθεση για τα σειρματόσκηνα. Να σα δώσω το λόγο. Thank you. Uh, oh, um, Ευχαριστώ. Α, να τα πω ισπανικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πολλούς γιατί είναι πολύ τεχνική η έκθεση και καταλαβαίνετε ότι χρειάστηκα πολύ μεγάλη βοήθεια και από τη Λούσια Άντερσον και από την Σαρανόβα και σας ευχαριστώ πολύ για τις συζητήσεις που είχαμε και θα ακολουθήσουν και άλλες για τις τροπολογίες. Η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κ. Δηλάου ήταν πολύτιμη και της κυρίας ε, Γκέρα που μας βοήθησαν πάρα πολύ για τα τεχνικά θέματα για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Ιδιαίτερα αυτό που ζητάει μια ομάδα συμφερόντων την οποία θα σας αναφέρω και θέλω να ευχαριστήσω και την Άστρη και τον Σεμπαστιάν στην γραμματεία. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, σε αυτά τα τεχνικά θέματα Υπάρχουν πολλές επιλογές κάθε φορά. Γι' αυτό έχουμε και 42 τροπολογίες, τις οποίες ήδη έχω συζητήσει με τους συντάκτες, τις υπόλοιπες αργότερα, στη συνεδρίαση που θα έχουμε με τους σκιώδες συγητές στις 24 Φεβρουαρίου. Θα ήθελα να τονίσω μερικές τροπολογίες ε, που θεωρώ σκόπιμο να συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Πρώτον, στις 3 Δεκεμβρίου συνεδριάσαμε και έκανα αυτή την ε, έκθεση και παρουσίασα. Η στρατηγική θα πρέπει να είναι κοινή για το νέο νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της αγοράς. Μετά από τη συνεδρίαση αυτή πρότεινα αυτές τις ε, ε, εκθέσεις και στη Βίκη Φόρ, την πρόεδρό μας, και στην Κάθριν Στάιλερ, αλλά και στους και οδησίγητες για τις εγκαταστάσεις ε, μεταφοράς με σειρματόσχηνα για να δούμε τι γίνεται με τις εκτελεστικές πράξεις, implementing act. Όπως γνωρίζετε αυτή η διαδικασία ήταν θέματα που αμφισβητήθηκαν επίμαχα, ιδιαίτερα ε, για να τα βρουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Συμβούλιο. Και η νομική μας υπηρεσία ε, εξέφρασε επιφυλάξεις ε, τις τροπολογίες 79 και 80 τις έχω αποσύρει και η Ντίτα και η Λούση και η Κάθριν ε, έχουν επιβεβαιώσει αυτή τη δράση και τις τροπολογίες οπότε νομίζω ότι έχουμε κοινή προσέγγιση. Δεύτερον, μια γαλλική ομάδα συμφερόντων μας επισήμανε και μάθαμε ότι υπάρχει ένα θέμα με τα φρένα αυτών των εγκαταστάσεων με τα σηματόσχηνα. Είναι οικονομικό και πολιτικό το θέμα γιατί λέγουν ότι η παρούσα διατύπωση του κανονισμού αποτρέπει την τεχνολογική ανάπτυξη μιας εταιρείας και εκείνοι λέγουν, ισχυρίζονται ότι ευνοεί άλλες εταιρείες με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ευχαριστώ πολύ γιατί ήταν πολύ περίπλοκο το θέμα. Καταλήξαμε σε ένα κείμενο που σέβεται την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και επιτρέπει σε όλες τις εταιρείες να αναπτύξουν τις τεχνολογίες τους και να έχουν ανταγωνισμό. 183 είναι η τροπολογία και την έκανα μαζί με την Τίτα Σάρας Νόβα. Υπάρχει και άλλη τροπολογία των Φελίπ Ζουάν και Νταντάν, των Γάλλων συναδέλφων, που νομίζω ότι απουσιάζουν αυτή τη στιγμή, αλλά φυσικά θα το συζητήσω μαζί τους αν χρειαστεί να φτάσουμε στη συμβιβαστική τροπολογία. Υπό την προϋπόθεση όμως, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, ότι θα υπάρξει τεχνολογική ουδετερότητα εγγυημένη. Η σκιώδηση συγκήτρια Λούση Άντερσον έχει κάνει περίπου τις μισές τροπολογίες Είχα την ευκαιρία να την ευχαριστήσω και να το συζητήσω ε, έτσι, επί της ουσίας μαζί της και θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα κάποιες τροπολογίες που ζητούν μεγαλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, παραπέμπει στην ιστοσελίδα του προϊόντος όταν είναι δυνατό αυτό και τη δήλωση συμμόρφωσης ε, στο άρθρο 3 ε, με τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, ενδιαφέρον είναι αυτό, αλλά θέλω να ακούσω και την άποψη Ευρωπαϊκής επιτροπή σχετικά. Μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας. Σε... Περιμένω ενδιαφέρον να ακούσω τα σχόλιά σας, διευκρινήσεις για τις τροπολογίες για να το σημειώσω και να προετοιμάσω την συνεδρίαση των σκιωδών, όπως σας είπα θα λάβει χώρα στις 24 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Thank you. Lucy Anderson. Ευχαριστούμε Λούση Άντρισον για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ όλους εδώ για τη δουλειά τους, ιδίως τον εισηγητή που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά για να συνδυαστούν όλα τα στοιχεία του. Δεν ήταν απλό, γιατί μερικά τα τεχνικά και νομικά θέματα και με πιέσεις από λομπίστες, όπως εξόγησε ο Αντώνιο, Αντώνιο έπρεπε να συναρθρωθούν ε, Πάντως καλύπτονται πολλές από τις ανησυχίες μας. Τα ζητήματα που ανέφερε τα εξέθεσε πολύ σωστά, δεν χρειάζεται να προσθέσω πολλά. Απλώς μια συνολική επισκόπηση. Οι τροπολογίες που, βάλαμε εμείς, όπως η αρχή της προφύλαξης, για την διευκρίνηση του ορισμού των τελικών χρηστών των σωματοσκήνων και ποιε είναι εδώ οι απόψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνουν κάποιες αλλαγές θέλαμε στο κείμενο για να αντικατοπτριστούν οι απαιτήσει για την ασφάλεια των ε, χρηστών και του σχετικού κειμένου με πρόσθετο βαθμό προστασίας. Συνυπογράψαμε τις τροπολογίες που εξαλείφουν τις αναφορές της ε, εφαρμοστικές πράξεις. Και οι τροπολογίες 138-183 για τον συμβαστικό ορισμό μας βρίσκουν θετικούς. Βεβαίω θα πρέπει να δούμε όλο τον κατάλογο των προτινόμενων αλλαγών, αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε επιτελέσει πρόοδο. Δεν μπορώ να πω ότι απαραίτητο θα συμφωνήσουμε με όλα, όλε τι τροπολογίε των άλλων συναδέλφων που είδαμε μόλι πρόσφατα, αλλά έχουμε χρόνο για αυτά τι ερχόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ. Ντάνι εκπροσωπεί την αίμα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, εκπροσωπώ, γιατί δεν μπορεί να έρθει. Εμείς οι συντηρητικοί υποστηρίζουμε τις περισσότερες από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και των σκιωδών και της εισηγήτριας, γιατί το κείμενο συμφωνεί και με τον κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. εκτός από τα θέματα που καλύτερα θα ήταν να καλύπτονται από εθνική νομοθεσία, όπως ορισμένα ανταλλακτικά. Γιατί το να καλυφθούν και αυτά από τον κανονισμό θα αύξανε το κόστος γενικότερα το κόστος. Αλλά γενικά οι συντηρητικοί στηρίζουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, δύο θέματα με ενδιέφεραν και εγώ υποστηρίζω την εξαίρεση, αλλά το πρώτο θέμα ήταν η εποπτεία της αγοράς και η διασφάλιση του ότι αυτό θα συμμορφώνεται με, τη μελλοντική, με το μελλοντικό κανονισμό εποπτείας της αγοράς. Είμαι ικανοποιημένη από την εισήγηση και ό,τι λέει. Μερικές από τις τροπολογίες μας όμως μπορεί να, μερικές από τις τροπολογίες μπορεί να θέσουν προβλήματα για μένα. Είναι τεχνικό το θέμα που αφορά την ασφάλεια, κανόνες ασφαλείας. Και πρέπει να είναι τεχνολογικός ουδέτεροι να μην προωθούνται ιδιαίτερα ορισμένες χώρες ή ορισμένη παραγωγή, είτε είναι Γάλλοι είτε η Γερμανία. Οι συμβιβασμοί που μπορεί να γίνουν στις τροπολογίες και μπορεί να καταλήξουν στην απώλεια αυτού του δέτερου χαρακτήρα θα ήταν κάτι αρνητικό. Θα διασφαλίσω λοιπόν με τον εισηγητή ότι θα ωφελεί όλους τους καταναλωτές και παραγωγούς. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω στα ισπανικά τον συνάδελφο εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Πασκάλ απουσιάζει. Ήταν η τελευταία ομιλήτρια. Α, η Ρόζα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Αντώνιο για την εξαιρετική του δουλειά. Ίσως δύο λόγια στα πολωνικά Συμφωνώ κι εγώ ε, και πρέπει να πω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ κέρια. Η απλούστευση κάποιων κανόνων, η διευκρίνηση κάποιων ρυθμίσεων που δεν ήταν ε, σαφής στην προηγούμενη οδηγία, ιδίω. για τις διαδικασίες που θα υλοποιούνται, αυτά είναι πολύ σημαντικά. Εγώ είχα προτείνει όμως και άλλα δύο σημεία που τα θεωρώ σημαντικά. Για τις χειμερινές αθλητικές δραστηριότητες, αυτές θα αλλάξουν πολύ, οπότε πρέπει να επεκτείνουμε την, τον ορισμό της οδηγίας των ορισμών για, τα, για, τα, για τις εγκαταστάσεις με σερματόσκηνα. Με, όχι, να μην το περιορίσουμε μόνο στο σκι δηλαδή ή στα snowboard. Πρέπει να διευρυνθεί ο ορισμός για όλες τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για αθλητικούς και τουριστικούς σκοπούς. Όλες δηλαδή οι νέες εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιήσουμε άμεσα ή στο αγγίς μέλλον. Επίσης η στο αγγισιο μελλον σιδηροδρομικών γραμμών. Ε, μην περιπλέξουμε πολύ το θέμα εδώ ούτε τις διαδικασίες ε, έγκρισης και πιστοποίησης. Γι' αυτό έχω αποβάλει την δική μου τροπολογία για να υπάρχει και κάποια διαβεβαίωση ότι στο μέλλον μπορούμε να φτιάξουμε καταστάσεις βάσει μια αίτηση, μπορεί κανεί να φτιάξει εγκαταστάσει, βάσει μια μιας αίτηση προ του ε, φορεί τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα ήταν μια πρόταση που θα μπορούσε να καλύψει τι ανάγκες μας. Ευχαριστούμε. Αντώνιο, θέλεις πάλι το λόγο. Έχει σχόλια να προσθέσεις κάτι σε αυτά που πάνε οι συνάδελφοι. Yeah, thank you. Uh, uh, Ευχαριστώ τη Λούση για αυτήν την ε, θετική προσέγγιση προς την τροπολογία 183. Δεν είναι απλό, αλλά το λαμβάνω υπόψη και Είμαι βέβαιο ότι τι τροπολογίε θα τι ξανασυζητήσουμε στι 24 με λεπτομέρειε. Για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστές, τα ιστορικά α, είναι εκτό. Υπάρχει μια τροπολογία από την δική μου ομάδα. Φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε για τα ιστορικά απελευθερή και το ίδιο και για τον συνάδελφο από του φιλελεύθερου για το θέμα των ιστορικών περιπτώσεων και παρακολούθηση τη αγορά. Αναμένουμε τι σχετικέ συζητήσει για την οδηγία, αλλά θα ήθελα να ε, αναφερθεί και να προσαρμοστούμε και στις μελλοντικέ ανάγκες. Για την τεχνολογική ουδετερότητα, βεβαίω, το είπα και στη δήλωσή μου. θα υπάρξουν συνεννοήσεις με το τι θέλουν οι μεν και οι δε, όπως με τους Γάλλους συναδέλφους, γιατί για μένα είναι κόκκινη γραμμή η τεχνολογική οδετερότητα στις συνομιλίες μου μαζί τους και τις λεπτομέρειες, όπως είπε και ο φίλος από τους Πασίνους, οι φίλοι από τους Πασίνους για, για τον αθλητισμό, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με το πεδίο. Τα όρια αφορούν τι εγκαταστάσει που επηρεάζονται και το τι θέλουμε να πετύχουμε με τους κανόνες μας. Αλλά είμαι ανοιχτό. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε στις 24. Πρόεδρε, θα ήθελα και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Γιατί Έχω θέσει κάποια ερωτήματα. Ιδίω για τον ορισμό. Ήθελα την άποψή σα εδώ. Γιατί απασχολεί και μερικού από του συναδέλφου. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλετε το λόγο για το θέμα των ορισμών. Ε, so, uh... Ευχαριστώ. Μπορούμε να υποβάλουμε σχόλια για τις τροπολογίες. Ε, Συντόμως. Α, συντόμως, λοιπόν. Πολύ συντόμως. Υπάρχουν, σας ευχαριστώ καταρχήν για τις τροπολογίες, μερικές από αυτές θέτουν, μας θέτουν προβλήματα. Όπως για την εισαγωγή της ρήτρας φρόνησης, διότι εδώ πρόκειται για κανονισμό όπου δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Άρα η, γιατί η ρήτρα φρόνηση εδώ εμπεριέχεται ήδη. Η σύγχυση είναι ότι όλες οι ρήτρες είναι δεσμευτικές και οι εποπτικές αρχές της αγοράς μπορούν να γνωρίζουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη ρήτρα αυτή της φρόνησης. Τώρα για τον ορισμό πιστεύω ότι αφορά, αναφέρεται στο document of conformity. Αλλά αυτό δεν είναι ορισμός που έχει εκεί μέσα. Είναι κανόνες. Κανόνες που είναι ήδη στα σημεία και στην προσθήκη στο παράρτημα. Και άρα όλα είναι το θέμα του declaration of conformity που λέμε. Ε, θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε την τροπολογία 153 όπου θέλουμε να παραμείνει το κείμενο ως είχε διότι η τροπολογία 153 παραλείπει, διαγράφει ορισμένες φράσεις. Η 155 εμπεριέχεται ήδη στα άρθρα στα σημεία 41 και 43, δεν χρειάζεται λοιπόν. Γενικές αναφορές στον τουρισμό και σε αθλητικές εγκαταστάσεις επίσης εμπεριέχονται, άρα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο κανονισμός αυτός γενικά respect to what is covered uh, by the regulation uh, αφορά μεταφορές βασικά, μεταφορές συγκοινωνίες, transporting function και στην 173 στην επίσης υπάρχει πρόβλημα. Αφορά τη θάλασσα. Εδώ αυτό που θέλουμε είναι να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση πυρκαγιάς σε τελεφερίκ και αυτό τίθεται μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς και άρα ισχύουν οι στάνταρ κανονισμοί. Εμείς προτιμούμε την 183 Αν χρειαστεί μπορούμε να κάνουμε αναφορά στα συγκεκριμένα οχήματα αλλά είπαμε ότι η τεχνολογική ουδετερότης πρέπει να διαφαλίζεται εδώ. Αν θέλετε κι άλλα, να σας πω κι άλλα. Ευχαριστώ. Thank you for that clarification. Thank you to everyone for their work on this. Ευχαριστώ όλους για τη δουλειά τους επί του θέματος. Θα ψηφίσουμε στις 17 Μαρτίου στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, ίδια ημέρα που θα ψηφίσουμε παρόμοιο χρονοδιάγραμμα. τα τρία θέματα που έχετε αναλάβει εσείς, εγώ και η Κάθριν. Αυτά θα καταλήξουν κάπου τον Ιούνιο, αλλά όταν υπάρχουν παρόμοια θέματα μπορούν μερικές φορές να συνδυαστούν και στους τριμερείς διαλόγους. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την έγκαιρη προετοιμασία και ιδίω για θέματα παρακολουθήσης τη αγορά και όλα αυτά. Ναι, μπορούμε να το δούμε μαζί. Εσείς είσαστε λοιπόν ο, ο επικεφαλής μας εδώ. Επόμενο σημείο στην εμερήσια διάταξη, αναθεώρηση του πλαισίου για την ε, διακυβέρνηση με σχέδιο γνωμοδότησης ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, όπου η συγκεντρία είναι ο συνάδελφος Μπερές. Και δική μας εισηγήτρια, κυρία Καλπέλτ. Παρακαλώ, αυτό το λόγο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω το σχέδιο αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε αυτό το θέμα. Το έχουμε ξαναδεί με τους σχεδόν ηγητές. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζω να κατάφερα να συμπεριλάβω και τις δικές σας απόψεις στη γνωμοδότησή μου. Βεβαίω γνωμοδότηση είναι. Δεν έχουμε ούτε χώρο ούτε χρόνο πια. Θα ήθελα όμως οπωσδήποτε να τονίσω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να σας εξηγήσω γιατί επέλεξα τη συγκεκριμένη ε, δομή και τι στοχεύω. Τι έδειξε η κρίση, ότι στα διάφορα κράτη-μέλη ε, ήταν διαφορετικές οι αντιδράσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να βρούμε ε, όλοι μαζί έναν τρόπο για να επιτύχουμε τους σκοπούς μας, που είναι κοινοί οι στόχοι. Ας πούμε, πώς θα ε, ενισχυθεί η διακυβέρνηση οικονομική και πώς θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Γνωρίζουν οι συνάδελφοι, δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί το θέμα, υπήρξε και προηγουμένως έκθεση σχετική και γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να μην βάλουμε όλα τα θέματα και στις δύο εκθέσεις. Δεν θα πρέπει να επαναλαμβανόμαστε, γνωμοδότηση είναι αυτό επαναλαμβάνω. Ποιο είναι το υπόβαθρο για την γνωμοδότηση αυτή ένα νέο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική διακυβέρνηση που παρουσιάστηκε στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Και εκεί αναφέρονται δύο θέματα. Πρώτον, η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και μια ευρωπαϊκή εποπτεία, όπως οι προτεραιότητες της Ευρώπης 2020 και οι στόχοι του προγράμματος αυτού. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι η διατήρηση της ε, σταθερότητας της Ευρωζώνης. Νομίζω λοιπόν ότι στη δική μας γνωμοδότηση θα πρέπει να εστιάσουμε την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι το θέμα μας. Και εκεί να κάνουμε προτάσεις. Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό μας αφορά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Θα ήθελα να προτείνω το εξής για να μπορούμε να συζητούμε για πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη εποπτεία της εσωτερικής αγοράς. Και θα πρέπει να βρούμε το σωστό και καλό πλαίσιο για να γίνει αυτό. Και εντός του πλαισίου αυτού να κινούμαστε και να βλέπουμε τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα των πολιτικών που ασκούν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια καταγραφή της κατάστασης αρχικά ε, και αυτό θα οδηγήσει σε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Από εκεί και πέρα θα έχουμε μια συνολική εικόνα την οποία θα μπορούμε να βελτιώσουμε. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την παρακαλέσω κάθε χρόνο να καταθέτει μια έκθεση για την πρόοδο στο πλαίσιο αυτό της εσωτερικής αγοράς, την οποία θα παρακολουθεί και παρακαλώ τους συναδέλφους να με υποστηρίξουν σε αυτή μου την προσπάθεια. Είμαι βαθύτατα πεπισμένη ότι ε, αυτή η παρακολούθηση της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να ακολουθεί το ευρωπαϊκό εξάμεινο και μάλιστα να ενταχθεί και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Είναι αλληλένδετα αυτά. Γι' αυτό μιλώ για ετήσια έκθεση. Κάθε χρόνο να καταγράφουμε, να κάνουμε μια φωτογραφία ας πούμε, της κατάστασης. Ε, προχωρήσαμε, υποχωρήσαμε για να υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο και μια πλατφόρμα που να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους μας. Και απαραίτητο. Ε, στην γνωμοδότησή μου αναφέρομαι και στη λογοδοσία, την υποχρεωτική και το δημοκρατικό έλεγχο και επίσης λέγω στη γνωμοδότηση ότι με τα μέτρα αυτά και την ευθύνη των κρατών μελών θα είμαστε τελικά σε θέση να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά και να την κάνουμε πιο διαφανή. να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι τα εμπόδια για να τα καταργήσουμε και να έχουμε ακόμα πιο αποτελεσματική δράση σε ό,τι αφορά τις τέσσερις ελευθερίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Α, και με χαρά περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας. Νίκολα Ντάντη. Ε, Νίκολα Ντάντε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που υπέβαλε ένα σχέδιο γνωμοδότησης πολύ καλά ε, Συμφωνούμε σε πολλά σημεία. Απλώς μερικές παρατηρήσεις για όσα ακούστηκαν και μερικές προτάσεις τις οποίες θα, φροντίσουμε να τις διευκρινίσουμε στη συνέχεια τη συζήτηση και με τι στενέ συνομιλίε που έχουμε με την εισηγήτρια και την οποία ούτω ή άλλω ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή έρχεται σε ένα χρονικό σημείο σημαντικό. Ε, έχουμε μπροστά μα μια περίοδο που οι κανόνε με τι πρώτε πράξει τη επίτροπή έχουν ε, ερμηνευτεί με διαφορετικού τρόπου σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη φάση μα έχει θέσει τρει πρωταρχικού στόχου. Την ανακοίνωση της για τις επενδύσεις, την ανακοίνωση για την ευελιξία. Να κινητοποιηθούν κονδύλια για τις επενδύσεις, να διασυνδεθούν οι επενδύσεις με την πραγματική οικονομία και να βελτιωθεί το ε, πλαίσιο για τις επενδύσεις. Πιστεύω ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα οικονομική διακυβέρνηση όπως έχει ονομαστεί, πρέπει αυτούς τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρώτες τη πράξη να τους συμπεριλάβουμε στους πρώτους μήνες εργασίας. Αυτό σωστά διευκρινίζεται στο σχέδιο γνωμοδότησης, στο σχέδιο έκθεσης. Γνωμοδότησης μάλλον, που η συγγήτρια έχει ετοιμάσει και είναι μια ευκαιρία για να συνδυάσουμε και πάλι την ε, οικονομική διακυβέρνηση με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Έχουμε πολλές φορές παρα, παρα, παρακολουθήσει να υπάρχει απόσταση μεταξύ οικονομικής διακυβέρνησης και πραγματικής οικονομίας. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτού του πρώτου μήνε εργασία τη έχει θέσει και πάλι στο επίκεντρο των ενδιαφέροντό τη το θέμα αυτό και θα πρέπει, έχοντα την αρμοδιότητα τη εσωτερική αγορά, ε, να ξανασυνδυάσουμε την οικονομική διακυβέρνηση με την εσωτερική αγορά για τι ανάγκε τη. Γι' αυτό στηρίζουμε και συμμεριζόμαστε την πρόταση που μα έχει υποβάλει η το σχέδιο γνωμοδότησης. Να υπάρξει και πάλι ετήσια αποβολή ε, έκθεσης για την εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς ε, χάρη στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμένου με συγκεκριμένε συστάσεις προς τα κράτη ανατομέα. Είναι μια αριστή πρόταση και τη στηρίζουμε. Υπό την οπτική γωνία της συνεργασίας να υπογραμμίσω κάποια σημεία. Πρώτον, το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια τέλεια ευκαιρία για να ε, εξελιχθεί η εσωτερική αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι στη νέα οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς που μπορεί να επιτρέψει πραγματική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στο διεθνές προσκήνιο για την Επιρό μας. Επίσης, να πω πως μέρος των επενδύσεων μπορούν να στοχεύσουν να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η ενιαία αγορά. Σκέφτομαι το θέμα του, της ψηφιακής ατζέντα, των υποδομών μεταφορών και υπηρεσιών, τη στήριξη των ευθύνων επιχειρήσεων, την ε, επαναμηχανήση. Αυτά είναι θέματα όπου οι επενδύσεις μπορούν να συμβάλλουν και η νέα ευρωπαϊκή διακυβέρνηση να είναι ένα σημείο συνδυασμού της πραγματικής οικονομίας με τη χρηματοπιστωτική και τις κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης. Η άλλη μου παρατήρηση είναι ότι η ρήτρα για τι επενδύσει, όπω την ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή τη για την απελευθερία, θα μπορούσε να μα οδηγήσει να προβλέψουμε και να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι η εσωτερική αγορά εφόσον υπάρχουν στοχευμένε επενδύσει από δημόσιου φορεί και όχι μόνον, θα μπορούσε λοιπόν να υποφεληθεί από του κανόνε ευελιξία που προέβλεψε στην ανακοίνωσή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν τέλει, πιστεύω και θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η συγγήτρια στην προηγούμενη παρέμβασή τη, ότι υπό το πρίσμα τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, για το 2020 είναι πολύ σημαντικό να δοθεί και πάλι να επανέλθει το κέντρο βάρους στην πραγματική οικονομία και το συνδυασμό της με την ε, εσωτερική αγορά και τις ανάγκες της και την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό για την Ευρώπη του 2020 και τη στρατηγική τη, αλλά και ένα από του κεντρικού πυλώνε όπου εμεί η Επιτροπή Προστασία των Καταναλωτών και Εσωτερική Αγορά μπορούμε να συνεισφέρουμε για να ενισχυθεί αυτή η εσωτερική αγορά. Είμαστε στη διάθεσή σα, είμαι στη διάθεσή σα για να συνεννοηθώ μαζί σα η συγκήτρια, αλλά και με του υπόλοιπου και και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ένα σημείο συμφωνίας που να ικανοποιήσει από την πολύ καλή ούτως ή άλλως ε, αφετηρία που ξεκίνησε στη δουλειά της εισηγήτρια να οδηγήσουμε σε μια χρήσιμη συνεισφορά στην Επιτροπή μας ε, για να εκφραστεί σωστά και η δική μας η θέση. Σε ευχαριστούμε Νίκολα. πάρα πολύ τον εισηγητή πάλι για την εξαιρετικά σκληρή του εργασία για να διασφαλίσει ότι θα τονίσουμε ιδιαίτερα τη διάσταση της ενιαίας αγοράς. Εδώ τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να βγάλουμε όλες τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς, να τις ξεκλειδώσουμε ώστε να καταλήξουμε σε απασχόληση, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, κέρδη. Και επίσης γνωρίζουμε ότι συχνά υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ ανάληψης πρωτοβουλίας και εφαρμογής της. Και από ό,τι κατάλαβα, ο στόχος είναι να δούμε εάν και κατά πόσον με τον ετήσιο κύκλο της εποπτείας της διακυβέρνησης μπορούμε να εξετάσουμε και τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Αλλά βέβαια η αγορά αφορά τις αγορές και τους καταναλωτές, ενώ η οικονομική γενικότερη διακυβέρνηση αφορά συνήθως δημόσιες δαπάνες και όχι τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς θέλουμε να δούμε αν τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για... με καθυστέρηση ή όχι. Ένα παράδειγμα η οδηγία των υπηρεσιών από το 12 ήδη είχαμε πει ότι θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε σχεδόν ένα πρόσθετο εκατοστιαίο σημείο ανάπτυξης, ίσως και παραπάνω, με μόνο αυτή την οδηγία. Γιατί λοιπόν δεν εφαρμόζονται τέτοια πράγματα ως τμήμα της γενικότερης οικονομικής διακυβέρνησης. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσουμε το θέμα της εφαρμογής, εφαρμογής της ενιαίας αγοράς. Γιατί εκεί μπορούν τα κράτη-μέλη να έχουν αποτέλεσμα. Όταν δέχονται μία νομοθεσία που αφορά την εσωτερική αγορά να την εφαρμόζουν και όλα. Και αν όχι να εξηγούν γιατί. Λοιπόν, στο τμήμα 6 της έκθεσής σας εγώ θα μιλούσα για ετήσια έκθεση εφαρμογής της ενιαίας αγοράς, όχι όπως το είπατε εσείς. Να λέμε δηλαδή γιατί δεν τα εφαρμόσατε αυτά και η Κομισιόν μας είπε στο πρόγραμμα εργασιών της ότι υπάρχει θέμα εφαρμογής που είναι και μάλιστα και το κλειδί, το κλειδί. Τώρα για το σημείο 4 κάτι σύντομο. πρέπει να τονιστεί ότι η οικονομική διακυβέρνηση είναι εταιρική σχέση μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Ο... Καλύτερη εφαρμογή κτλ. Να προσέξουμε δηλαδή στις διαβουλεύσεις να μην περιοριστούμε σε επενδεδημένα συμφέροντα. Γιατί είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι. Να βάλουμε λοιπόν μια διατύπωση που να λέει ότι είναι η διαβούλευση αλλά χωρίς να χάσουμε την ανεξαρτησία. Την ανεξαρτησία λέγω τέλεια. Αυτά είναι οι σκέψεις μου και προσβλέπω και εγώ στη συνεργασία σας. Ευχαριστώ. Η Ούλα τώρα, η Ούλα από τους Ελεύθερους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ την Ισογετρία για την πολύ καλή δουλειά, για την γνωμοδότηση αυτή. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η εσωτερική αγορά είναι ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο μόνος τρόπος να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Αυτό σωστά το είπε και η Πρόεδρος και οι περισσότεροι στην ε, παρέμβασή τους. Γι' αυτό λοιπόν βασικό μας καθήκον είναι να δούμε Πώ θα λειτουργήσει καλύτερα η εσωτερική αγορά συνδυασμό με την οικονομική διακυβέρνηση. Νομίζω η γνωμοδότηση ΙΜΚΟ θα προσφέρει μια πολύτιμη συνεισφορά για την έκθεση τη Επιτροπαϊκής Οικονομικών Υποθέσεων όπω και η γνωμοδότηση τη Επιτροπή απασχόληση. Θα μα προσφέρει και μια άλλη οπτική γωνία για το θέμα. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να τονίσω ορισμένα σημεία που μα ενδιαφέρουν ε, ως το σχέδιο που έχουμε μπροστά μα Πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει να μείνουμε στην πορεία της μεταρρύθμισης. Άκουσα ορισμένους να λένε ότι ίσως υπάρξουν δυνατότητες να προβλεφθεί ευελιξία για το δημοσιονομικό πλαίσιο, για να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη. Όμω δεν είναι αυτό ο τρόπο να προχωρήσουμε, όπω το βλέπω εγώ. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε τώρα του κανόνε. Οι μεταρρυθμίσει φέρνουν αποτελέσματα. Τα ελλείμματα μειώνονται. Και η Ευρώπη πολύ αργά αλλά αποτελεσματικά ανακάμπτει. Πρέπει να συμμορφωθούν περισσότερο οι χώρε με τι αναχώρα συστάσει. Η οικονομική διακυβέρνηση δεν θα έχει καμία αξία αν τα κράτη-μέλη δεν ακολουθήσουν τι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα τρόπο για να υπάρξει καλύτερη συμμόρφωση θα είναι να υπάρξει αναλήψη ευθύνη από τα εθνικά κοινοβούλια για τι αναχώρα συστάσει. Μια άλλη πρόταση είναι να διασυνδέσουμε την πρόσβαση με την στήριξη από το επενδυτικό πρόγραμμα και την συμμόρφωση προς τις συστάσεις. της Επιτροπής. Ίσως αυτό να υπάρξει, να ακουστεί αφιλεγόμενο, αλλά πιστεύω θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Επίσης θα έπρεπε να έχουμε μια σαφέστερη μνήμα προς την παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη σημασία τη, διότι έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση εδώ στην ενιαία αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Επίση, να επικεντρωθούμε στου τομεί τη εσωτερική αγορά που θα προσφέρουν περισσότερη πιστιθέμενη αξία. Όπω η ενιαία ψηφιακή αγορά που είναι μια ύψιστη προτεραιότητα για μας και όπου έχουμε ήδη πολύ καλές συζητήσεις για μέρη της πρότασης. Αυτές, αυτά είναι τα σχόλιά μου σε αυτή τη φάση και αν υπομονώ να συνεργαστώ με την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Ο Ντένις αποσιάζει σήμερα. Είναι σκιώδης της Γκουε και από τους Πρασίνους ο Πασκάλ Τιουραν. Θες το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ πολύ γρήγορα γιατί περνάει χρόνος να ευχαριστήσω την κυρία την εισηγητρία για τη δουλειά της ε, και να επιμείνω στην ανάγκη να έχουμε μια πιο ενιαία προσέγγιση μέσα στο δυνατόν περισσότερο συμμετέχοντες και το Κοινοβουλίο σε ένα δραστήριο ρόλο. Ε, λοιπόν τις δικές σας προτεραιότητες και συμφωνούμε. Επί της ουσίας δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν θα καλύψουμε τώρα το θέμα και εγώ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ασχολούμαι με τα θέματα αυτά, Ο και ο εισηγητής, ήδη συζητούνται και, και αυτά. Οι συζητήσει για τις επιπτώσεις και το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι ένα πραγματικό θέμα. Εγώ α, επί της αρχής έχω μια ε, Πρώτα μια μέρη να εκφράσω για την λειτουργία τη εσωτερική αγορά και την διακυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι η Ευρώπη ξεφεύγει σε μια λογική πολύ πιο λογιστική. Δεν λαμβάνει υπόψη να επαρκώ τον ε, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για την εσωτερική αγορά, αυτό που έχει προσπαθήσει η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο στο παρελθόν συμπεριλαμβάνοντα τι δημόσιε προμήθειε σε πολλά θέματα, τα κοινωνικά κριτήρια, τα περιβαλλοντικά και το καθεξής. Το λέω κάθε φορά, αλλά είναι θέμα ισορροπία. Ε, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν λάβουμε υπόψη το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και αν δεν δούμε βραχυπρόθεσμα πώ θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του χρέου και των εγκλημάτων. Ίσως αυτά να μας ε, κάνουν να διαφωνούμε, αλλά είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να το αναφέρουμε, να το συζητήσουμε, να το εξετάσουμε, για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα γλιστρήσουμε σε μια λογική μπακαλίστικη της Ευρώπης, ε, τεχνοκρατική μόνο. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτή τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διάσταση. Αλλά είναι μια τεράστια συζήτηση που δεν μπορεί να γίνει αυτή την ώρα στο επίπεδο αυτή τη Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Άλλοι ή ε, να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Στην εισηγήτρια. Κυρία εισηγήτρια, θέλετε να ανακεφαλαιώσετε. Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, για τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις και προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ. Αλλά κοιτάξτε, μια σελίδα έχω. Δεν χωράει και πάρα πολλά πράγματα μια σελίδα δεν μπορούν να χωρέσουν σε μία σελίδα όλα αυτά που είπατε. Βεβαίως βελτιώνετε την γνωμοδότησή μου με αυτά που λέτε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Συμφωνώ ότι θα πρέπει η οικονομική διακυβέρνηση να συνδεθεί με τη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς με τρόπο ολοκληρωμένο και ενιαίο. Συμφωνώ επίσης αυτό που είπατε για το επενδυτικό σχέδιο Juncker και υποστηρίζω τη γνώμη της Προέδρου. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Πριν κάνουμε οποιαδήποτε νέα πρόταση, να δούμε ποιες προτάσεις ήδη έχουν γίνει. Οι οδηγίες ε, που έχουν ε, υιοθετηθεί ε, τίθενται επαρκώς σε ισχύ, έχουν μεταφερθεί όπως πρέπει και αν όχι γιατί. Αυτό ε, είναι που μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες που μετρούν αυτά τα θέματα και θα πρέπει να παρακολουθούμε την ε, εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, θα πρέπει να βλέπουν τους εαυτούς τους ως εταίρους. Όχι αναγκαστικούς εταίρους, αλλά διαβουλεύσεις με διαφάνεια, με συνεργασία σε επικοδομητικό πνεύμα. Δεν θα πρέπει να το αντιλαμβάνονται ως κάτι που τους επιβάλλεται. Οι συστάσεις χώρα, για παράδειγμα, είναι κάτι που υποστηρίζουν τα ίδια τα κράτη-μέλη, εκπονούνται από κοινού. Γι' αυτό και τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν εδώ να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ε, εννοώ το δημοκρατικό έλεγχο που ασκούν στην εκτελεστική εξουσία. Ε, συμφωνώ για τις μικρομεσαίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι μάλιστα και η σπονδυλική στήλη, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Γι' αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που να οδηγούν σε ανάπτυξη. Δυστυχώς όμως στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Οι συστάσεις αναχώρα κινούνται ω προ την εφαρμογή του σε ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, μόλις 10%. Τι γίνεται αυτό. Πολλά κράτη-μέλη απλούστατα ε, δεν αποδέχονται πλήρως τις συστάσεις που τους γίνονται. Θα πρέπει να απευθύνουμε συστάσεις στα κράτη που να αντιπροσωπεύουν ε, ε, τους στόχους μας και να μπορούν να μετρηθούν αλλά και να υλοποιούνται τι να τις κάνω τις συστάσεις ανά χώρα αν δεν τις εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει ο καθής να αναλάβει τις ευθύνες του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις που εκδίδει, αλλά και τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να τα εστερνίζονται και να τα εφαρμόζουν. Και αν δεν τα εφαρμόζουν, να προτείνουν ισοδύναμα. Εναλλακτικέ προτάσεις δηλαδή. Είναι αδιαφυσβήτητη η σημασία των μικρομεσαίων για την ε, ψηφιακή αγορά. Ήθελα ε, κάπως να περιορίσω τη γνωμοδότησή μου και να την διαφοροποιήσω από την προηγούμενη έκθεση. Αν θέλετε να επαναλάβουμε τα όσα έλεγε η παλαιότερη έκθεση, τι να κάνω. Ο κύριος Πασκάλ Τζιρό έχει απόλυτος δίκιο. Η εσωτερική αγορά ε, είναι κάτι που δεν μπορεί να έχει στόχους βραχυπρόθεσμους. Θα πρέπει να έχουμε ένα μακρύτερο χρονικό ορίζοντα στην εφαρμογή όλων αυτών, με ισορροπία, αλλά οι πάντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υλοποιούν. Ε, με θετικές προτάσεις. Δεν είναι καταναγκαστική αυτή η προσπάθεια με το στανιό. Είναι αμοιβαία, υποφελής, εθελοντική βάση και ε, καλοπροαίρετα. Όλα αυτά θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω στη γνωμοδότησή μου. Φαντάζομαι θα κάνετε και εσείς τροπολογίες θα κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε η γνωμοδότηση αυτή να γνωρίσει όσο γίνεται μεγαλύτερη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 11 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Κοιτάξτε όλοι να αποβάλλετε γρήγορα τι τροπολογίες. σα. Ευχαριστώ και πάλι για τη δουλειά σα. Αυτό είναι το τέλο τη συνεδρίασης για σήμερα. Απλώς ίσω κάτι να έπρεπε να αναφέρω. Είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να οργανώσει εκδήλωση για τον εορτασμό τη δεκαετία από τη δημιουργία των κέντρων καταναλωτών. Στο Κοινοβούλιο μαζί ήρθε να οργανωθεί, αλλά πρέπει να το δούμε σε σχέση με τα νέα μέτρα ασφαλεία που έχουν προβλεφθεί για το Κοινοβούλιο. Μόλι ξέρουμε περισσότερα θα σα ενημερώσουμε. Για την ώρα όλοι κοιτάζουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, ενώ το πρωτόκολλο ασφάλειας του Κοινοβουλίου αλλάζει.